colleghi, la sessione di... Αγαπητοί συνάδελφοι, η απογευματινή μας σύνοδος ξεκινάει με θέματα πολύ επίκαιρα. Το πρώτο θέμα αφορά την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης στην Αίγυπτο και τις προοπτικές για μια μετάβαση σε μια πραγματική δημοκρατία. Που, προοπτική που φαίνεται όλο και πιο απόμακρη την περασμένη Παρασκευή, όπως ξέρετε, λίγο πριν από την προεδρική εκλογή, ο Αιγυπτιακός στρατός κύκλωσε το κοινοβούλιο και εμπόδισε τους βουλευτές που πρόσφατα είχαν εκλεγεί να πάνε στην Βουλή. Ταυτόχρονα έχουμε και την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου που θεώρησε αντισυνταγματικές τις πρόσφατες ε, βουλευτικές εκλογές. Αυτή η απόφαση δίνει στις στρατιωτικές αρχές ε, εξουσίες σημαντικές και θα έχει σημαντικό ρόλο στο, στη σύνταξη του νέου συντάγματος. Η αντιπολίτευση κατηγορεί το στρατό ότι παρενέβη για να μην επιτρέψει στον Αμέτ Σαφίτ ε, να συμμετάσχει και μιλάει για πραξικόπημα. Δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών και οι δύο ε, υποψήφοι κραυγάζουν την νίκησαν. Ο στρατός λέει ότι θα αναγνωρίσει τον ε, εκλεγμένο πρόεδρο και θα αναλάβει τα καθήκοντά του ο πρόεδρος αυτός στις 30 Ιουνίου. Όμως η κατάσταση παραμένει πολύ ανησυχητική. Μετά τα τελευταία γεγονότα στο στην Αίγυπτο και τις προοπτικές για την δημοκρατική μετάβαση, ε, θέλουμε να συζητήσουμε με τον Ιγκ Μιγκαρέλη, ε, ο οποίος ε, είναι διευθυντής ε, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και υπεύθυνο για την περιοχή αυτή. Σας ευχαριστούμε κύριε Μιγκαρέλη για την διαθεσιμότητά σας. Πέστε μας τι άποψη έχει η υπηρεσία σας για την κατάσταση στην Αίγυπτο, ε, πρώτο ερώτημα που είναι και εύκολο, Ποια είναι τα πιθανά σενάρια που προβλέπονται από την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για τι επόμενε μέρε και τι επόμενε εβδομάδε, τι θέσει προβλέπετε ότι θα έχει ο υποψήφιο των αδερφών μουσουλμάνων, που από πολλού θεωρείται ο νικητή, ο πιο επικρατέστερο υποψήφιο, και τι θέση θα έχει η υπηρεσία σα στι σχέσει με την Αίγυπτο και ιδίω απέναντι στο Ανώτατο Συμβούλιο ε, των Ένοπλων Δυνάμεων και Ενγέννητου Στρατού. Σας δίνω πάρα αυτό το λόγο, κύριε Μικαρέλη, για 10 περίπου λεφτά για να κάνετε αυτή την παρέμβαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά που με προσκαλέσατε και που είμαι εδώ για να μοιραστούμε τους προβληματισμούς μας, για να ακούσουμε τα ερωτηματικά που υπάρχουν για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αίγυπτο και γενικά στον αραβικό κόσμο. Λοιπόν, εδώ και μία εβδομάδα συνέβησαν πολιτικές εξελίξεις στην Αίγυπτο. Υπάρχουν όμως τέσσερις πολιτικές εξελίξεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ε, καταρχάς, την περασμένη Πέμπτη είχαμε δύο αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου ε, και πολύ σημαντικές αποφάσεις με πολιτική διάσταση. Καταρχάς, το δικαστήριο αποφάσισε, το συνταγματικό δικαστήριο αποφάσισε ότι η υποψηφία του Αχμέτ Σαφίκ, ε, του πρώην ε, α, α, στρατιωτικού της αεροπορίας, ήταν έγκυρη. Του επέτρεψε λοιπόν να συμμετάσχει στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Ε, Παράλληλο, που του επέτρεπε να συμμετάσχει στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, το Σταγματικό Δικαστήριο θεώρησε ότι ο νόμος με βάση τον οποίο οργανώθηκε η ε, εκλογή της συνέλευσης του λαού και κυρίως του ενός τρίτου του ενός τρίτου των βουλευτών που εξελέγησαν ο καθένας μόνος του, όχι με βάση κάποιους εκλογικούς καταλόγους πολιτικών κομμάτων, το δικαστήριο θεώρησε ότι αυτός ο νόμος δεν ήταν σύμμορφος προς το Σύνταγμα. Επομένως, ακύρωσε τις εκλογές του συνόλου των βουλευτών στο κάτω σώμα της Βουλής, που είναι η, συνέλευση, η Λαϊκή Συνέλευση, το Σώμα του Λαού. Αυτή είναι η δεύτερη πολιτική απόφαση που νομίζω ότι είναι μεγάλης πολιτικής εμβέλειας και λήφθη την Πέμπτη. Εν συνεχεία. Το και την Κυριακή είχαμε το δεύτερο γύρο, γύρο των προεδρικών εκλογών και την Κυριακή το βράδυ είχαμε ένα συνταγματικό διάταγμα από το Συμβούλιο, το Συμβούλιο των ενόπλων δυνάμεων που λέει ότι διαλύεται η Βουλή, το Κοινοβούλιο και έδωσε την νομοθετική εξουσία στο Ανώτατο Συμβούλιο των Ενόπλων Δυνάμεων. Φυσικά αυτό δημιουργεί μια ιδιάζουσα κατάσταση. Τώρα, αν ε, διατρέξουμε τα τέσσερα γεγονότα το ένα μετά το άλλο για τις προεδρικές εκλογές. Με βάση τις ε, αρχικές πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας και υπογραμμίζω το προκαταρτικά αποτελέσματα που δεν είναι επίσημα ακόμα. Ο υποψήφιο των ε, αδερφών μουσουλμάνων Μωαμέτ Μορσή κέρδισε το δεύτερο γύρο με περίπου 52% των ψήφων. Όμως, ο αντίπαλός του ο Αχμέντ Σαφρίκ, ο υποψήφιος του στρατού, αμφισβητεί το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών. Και το επίσημα, τα επίσημα αποτελέσματα θα τα έχουμε σε δύο μέρες, 21 του μηνός, την Πέμπτη. Ο Μοαχμέτ Μορσί θεωρεί ότι κέρδισε με 52% των ψήφων, ο Αχμέτ Σαφίκα αμφισβητεί αυτό το αποτέλεσμα που είναι προκαταρτικό και την 5η στις 21 Ιουνίου θεωρούμε ότι θα έχουμε τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών αυτών. Με βάση αυτά που μας λένε οι παρατηρητές μας, ο δεύτερος γύρος των εκλογών έγινε μέσα σε συνθήκες σχετικής ηρεμίας, το οποίο σημαίνει ότι οι εκλογές δεν έγιναν μέσα σε ένα τέλειο κλίμα, ε, στην διοικητική προετοιμασία των εκλογών υπάρχουν κάποια υπήρξαν κάποια προβλήματα, υπήρξαν και κάποιες παρατυπίες που διαπιστώθηκαν, όμως το σύνολο αυτών των παρατυπιών και των ε, διοικητικών ανεπαρκειών δεν ε, μοιάζει να μπορεί να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα των εκλογών. Με άλλα λόγια, όποιες και αν είναι αυτές οι παρατυπίες που έλαβαν χώρα, δεν αμφισβητείται ότι ο Μουαχμέτ Μορσί ε, έχει ένα προβάδισμα σε σχέση με τον αντίπαλό του, τον Αχμέτ Σαθίκ. Όλες αυτές, επαναλαμβάνω, είναι εκτιμήσεις που μας αποστέλουν οι εμπειρογνώμονές μας ε, επιτόπου, αλλά αν μου λέγανε ε, υπογράψτε το αυτό με τη ζωή σας, θα έλεγα, ε όχι, δεν φτάνω μέχρι εκεί. Είναι εκτιμήσεις με βάση αυτά που μας λένε οι εμπειρογνώμονές, οι εμπειρογνώμονές μας. Σύνεση λοιπόν, περιμένουμε μέχρι την 5η 21 Ιουνίου για τα τελικά αποτελέσματα. Θέλω να πω τώρα δύο λόγια για ένα άλλο γεγονός που έλαβε χώρα. Κυριακή βράδυ. Το ΣΚΑΦ, η η ο στρατός υιοθέτησε ένα διάταγμα που μεταφέρει όλη την νομοθετική εξουσία τι ενόπλες, δυνάμει. Ε, δυνάμεις. Διαλύεται το κοινοβούλιο και οι στρατιωτικοί παίρνουν όλη την νομοθετική εξουσία. Πέραν αυτού, οι στρατιωτικοί λένε ότι αν η συντακτική συνέλευση που δημιουργήθηκε πριν από αρκετές εβδομάδες και που μέχρι στιγμής δεν ήταν σε θέση να δουλέψει σοβαρά, εάν αυτή η συντακτική συνέλευση δεν αρχίζει να εργάζεται πάρα αυτά, Εμεί, οι στρατιωτικοί θα υποδείξουμε μια τέτοια συνέλευση η οποία θα εργαστεί για την ε, σύνταξη ενός νέου συντάγματος. Οι στρατιωτικοί επίσης μας λένε ότι θα έχουν δικαίωμα βέτο επί του επόμενου συντάγματος. Δηλαδή, αν θεωρήσουν ότι ένα άρθρο του συντάγματος που θα προκύψει δεν είναι συμβατό με τα υπέρτατα συμφέροντα της χώρας όπως τα αντιλαμβάνονται εκείνοι, έχουν το δικαίωμα να βάλουν βέτο επί του άρθρου αυτού. Ακόμα και αν είμαστε πολύ προσεκτικοί, όπως κάνουν οι γραφειοκράτες πάντα, που είναι πολύ προσεκτικοί, δεν μιλάμε εδώ τώρα για δημοκρατία. Και αν θυμηθούμε τι λέγανε οι στρατιωτικοί μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουλίου του 2011, ε, λέγαν τότε σε όλους τους επισκέπτες οι στρατιωτικοί και μάλιστα το είπαν στον Παρόζο, στην Άστον και σε διάφορους άλλους, ότι ήταν αποφασισμένοι να μπουν στα στρατόπεδά τους πριν το Δεκέμβριο του 2011. Θυμηθείτε τι λέγανε λοιπόν τότε και ό,τι συμβαίνει σήμερα. Και αν τα συγκρίνουμε αυτά, αν συγκρίνουμε τις, την πολιτική πραγματικότητα και τις πρακτικές τους, τότε τίθενται πολλά ερωτήματα. Παρότι υπάρχουν πολλές, πολλά ερωτηματικά για το τι θα συμβεί τα, τις επόμενες εβδομάδες. Πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα καταρχάς ε, της Πέμπτης για τον Πρόεδρο. Ε, συνεχεία θα σχηματιστεί η κυβέρνηση, ο Πρόεδρος θα υποδείξει έναν ε, Πρωθυπουργό. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι τους επόμενους μήνες την νομοθετική εξουσία θα την έχουν στρατιωτική. Δεύτερον, οι στρατιωτικοί κρατάνε το δικαίωμα να υποδείξουν μία συντακτική συνέλευση και τρίτον, στρατιωτικοί έχουν το δικαίωμα να αμφισβητήσουν και να βάλουν βέτο για οποιοδήποτε άρθρο του συντάγματο που θα προκύψει που και που το θεωρούν μη συμβατό με τα υπέρτατα συμφέροντα τη χώρα. Για να το πω πολύ συνοπτικά, έχουμε σοβαρότατε ανησυχίε για την δημοκρατική μετάβαση τη Αίγυπτου. Επίσης, 13 Ιουνίου, την περασμένη εβδομάδα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης υιοθέτησε ένα διάταγμα που επιτρέπει σε στρατιωτικούς να συλλάβουν πολίτες, τότε πραγματικά διερωτώμεθα τι κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις θα έχει ένα τέτοιο ε, διάταγμα και για ποιο λόγο το πήραν. Και παρότι λοιπόν την, ε, την, το περασμένο Σαββατοκύριακο έγινε έγιναν οι τρίτες εκλογές, τρίτες κατά σειρά, που συνέβησαν μέσα σε ένα κλίμα ε, σχετικής ηρεμίας μετά από 60 χρόνια αυταρχικού καθεστώτος, παρότι χαιρόμαστε για το γεγονός ότι από εδώ και πέρα θα γίνονται στην Αίγυπτο σοβαρές εκλογές, παρόλα αυτά η στρατιωτική πήραν μια σειρά από αποφάσει, οι οποίες ήταν ανησυχητικέ, ανησυχητικέ για όλους τους δημοκράτες και για όλους όσους έχουν συμφέρον να υποστηρίξουν την δημοκρατική μετάβαση της Αιγύπτου. Τι μπορεί να κάνει απέναντι σε αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς, επαναλαμβάνουμε ότι υποστηρίζουμε με όλη μας τη δύναμη τη δημοκρατική μετάβαση της χώρας και ότι είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε ανεπιφύλακτα σε ένα διάλογο με τις ε, δημοκρατικά εκλεγμένες αρχές ε, δηλαδή, ελπίζουμε με τον πρόεδρο και με, το, με την κυβέρνηση που θα διορίσει. Δύο, θα πρέπει παρόλα αυτά να υπενθυμίσουμε στους στρατιωτικούς ότι είχαν υποσχεθεί να μεταφέρουν την εξουσία σε μη στρατιωτικούς πριν από το Δεκέμβριο που μας πέρασε. Αυτό όμως δεν θα συμβεί γιατί επί μήνες ακόμα θα έχουν ε, την εξουσία στα χέρια τους, την νομοθετική εξουσία. Τρίτον, θα πρέπει να επαγρυπνούμε ούτως ώστε η διαδικασία εκπώνησης του νέου ε, συντάγματος θα συμπεριλαμβάνει του περισσότερους νατούς φορεί και ενδιαφερόμενου. Όλα τα τμήματα της Αιγυπτιακή κοινωνίας και τελευταίο σημείο και θα σταματήσω σε αυτό, θα πρέπει να πιέσουμε τις Αιγυπτιακές αρχές να λάβουν μέτρα απαραίτητα ούτω ώστε να σταματήσει τώρα η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης και αυτό σημαίνει η συμφωνία και με το Δουνουτού και μετά από αυτή τη συμφωνία, εμείς θα είμαστε σε θέση ως Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσουμε μια μακροοικονομική βοήθεια. Αυτά με δύο λόγια, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την Αίγυπτο σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ποιοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Πρώτος ο κύριος Σαλαφράγκα. Τρεις, τρία λεπτά ο κάθε ομιλητής για να έχουμε και χρόνο για απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Μεγκαρέλη που εξ ονόματος της ε, Διπλωματικής Υπηρεσίας ήρθατε να συμμεριστείτε μαζί μα στα τελευταία γεγονότα τα οποία αφορούν την κατάσταση στην Αίγυπτο. Αναφερθήκατε στην αξιολόγηση που έκαναν οι βεπαΐοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό, μετά το δεύτερο γύρο των ε, προεδρικών εκλογών, λαμβάνοντα υπόψη το, το γεγονός ότι δεν προσεκλήθη να αποστείλει παρατηρητές για τις εκλογές η Ευρωπαϊκή Ένωση στρίκτου σένσου, θα είναι μια, είναι μια αποστολή επαϊόντων. Θα ήθελα να ξέρω πόσοι επαϊόντες συναποτελούν αυτή την αποστολή και ποια είναι η άποψη που έχουν οι άλλες αποστολές παρατηρητών, διεθνών παρατηρητών, που έχουν προσκληθεί να παρακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία και θα ήθελα να ρωτήσω, λαμβάνοντα υπόψη ότι το πλαίσιο το οποίο αναφέρατε σε σχέση με τα προσωρινά αποτελέσματα και όχι τα τελικά, είναι 52% για τον νικητή υποτίθεται αυτών των εκλογών. Τι θα γίνει, τι γίνεται όταν ο άλλος ε, υποψήφιος αμφισβητεί τα αποτελέσματα. Υπάρχει κάποιο σώμα το οποίο μπορεί να διευθετήσει τις διαφορές σε σχέση για παράδειγμα με το συνταγματικό δικαστήριο. Πώς επιλύεται μια τέτοια αμφισβήτηση, ένα τέτοιο θέμα. Η δεύτερη ερώτηση για το δεύτερο στοιχείο που μας παρουσιάσατε και που είναι η ακύρωση της ε, συντακτικής συνέλευσης για λόγους, ας το πω έτσι, ατυπ παρατυπιών όσον αφορά τις, τα ποσοστά για τους υποψηφίους σε σχέση με τα κόμματα. Το κανονικό είναι όταν ακυρώνεται κάποια συνέλευση να απευθύνεται έκκληση για τη διεξαγωγή νέων εκλογών σε ένα νέο νομικό πλαίσιο ώστε έτσι να μπορέσει να θεωρηθεί ασκόπιμο αυτό που πρέπει να γίνει έτσι και νόμιμο μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο δεν θεωρείτε εσείς ότι θα έπρεπε να συγκληθούν ε, ε, γενικές εκλογές. Κατανοώ ότι δεδομένης της ασάφειας και αβεβαιότητας για τις προεδρικές εκλογές και σε σχέση με τον προσδιορισμό ε, κυβέρνησης υπουργών και τα λοιπά. Είναι ανησυχητικό όμως για την σύνταξη του νέου συντάγματος να μην υπάρχει νομοθετική εξουσία που άμεσα να έχει εκλεγεί από τους πολίτες ώστε να προχωρήσει ακριβώς στη σύνταξη αυτής της ε, συνταγματικής χάρτας του συντάγματος. Θέλω να ξέρω την άποψή σας. Εφόσον θα έχει αντιμετωπιστεί αυτό το, ε, αυτή η αμφισβητή αμφισβήτησης δεν θα έπρεπε να συγκληθούν νομοθετικές νομικές εκλογές για να καλυφθεί το νομικό χάσμα, το νομικό κενό που υπάρχει και υπό ποιους όρους θα μπορούσε να γίνει αυτό. Αυτές τις αρμοδιότητες δηλαδή να τις αναλάβει το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο. Πώς γίνεται αυτό. Τρία λεπτά ο κύριος Γκόμες, κυρία μάλλον, για τρία λεπτά. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Μιγκαρέλη, λέει η κυρία Γκόμες, για την ενημέρωση. Πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ θλιμμένη για όσα συμβαίνουν στην Αίγυπτο, αλλά δεν με εξέπληξαν. Είχα είχα ε, συνοδεύσει τον πρόεδρο της Βουλής όταν έγινε το δημοψήφισμα τον Μάρτιο του 2011 και είδα πόσο ενθουσιασμένος ήταν ο κόσμος τότε. Αλλά όταν συναντήσαμε τις αρχές είδαμε ότι τα πράγματα δεν θα πήγαιναν καλά. Διότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα άφηναν τα πράγματα να ευοδοθούν. Και η άρνηση να υπάρξει μία ε, αποστολή παρατηρητών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αίγυπτο είχε κάποιο νόημα διότι ακριβώς δεν θέλανε ε, να παρατηρήσουν να, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Ήταν ένα, μια ένδειξη, σημαντική ένδειξη. Επίσης ε, έγιναν φρικτά πράγματα. Παραδείγματο χάρη ότι οι γυναίκες έπρεπε να κάνουν τεστ ε, ε, παρθενίας ε, γιατί συμμετείχαν σε, διαδηλώσει στις διαδηλώσεις και στι εκδηλώσει του Μαρτίου κτλ. Επίσης, στο ΣΥΝΑ είδαμε ότι έχουμε μαρτυρίες για επίσης ε, φρικαλαιότητες που έγιναν από τις ε, φυλές των Βεδουίνων και έγιναν και απαγωγές ε, και τι, τα λίτρα ήταν 6.000 δολάρια πριν από λίγο καιρό, τώρα έχουν φτάσει στα 60.000 και έχουμε βιασμούς, δολοφονίες, πωλήσει οργάνων έχουμε τεκμήρια, έχουμε αποδείξεις και αυτά είναι στοιχεία για τα οποία θα έπρεπε να διαμαρτυρηθούν αν μη τι άλλο οι στρατιωτικές αρχές του, της Αιγύπτου και δεν το κάνουν για αυτά που γίνονται στην, στο Σινά παραδείγματο χάρη δεν έπρεπε να κάνουμε κάτι λοιπόν οτιδήποτε είπε ο κύριος Μιγκαρέλη είναι σωστό αλλά θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λέδη Άστον πρέπει να τονίσουν με πιο απόλυτους όρους ε, την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πούμε αρκεί. Για την αξιολόγηση τώρα των εξελίξεων θα έλεγα ε, θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην ανάπτυξη η οποία θα στηρίζεται στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτό είναι πρωταρχική σημασία. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηρίξει κάτι τέτοιο. Έστω και αν δεν μπορεί να συνδιαλλαγεί απευθείας με την κυβέρνηση, εάν η κυβέρνηση δεν είναι δημοκρατική, είναι να βοηθήσει την κοινωνία των πολιτών. Thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μιγκαρέλη για τις ε, αναλύσεις ε, που κάνατε, αναλύσεις με τις οποίες συμφωνούμε απόλυτα και πραγματικά ε, όντως πρόκειται για μια τραγωδία. Είμαστε σε επαφή και με τους νέους, οι νέοι αποτελούν μια δύναμη, μια ελπίδα που τώρα έχουν χάσει την, το όραμά τους, ε, δεν ξέρουν τι θα γίνει, προς τα που πάνε. Τώρα για το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης, της δημοσιονομικής ενίσχυσης. Ρωτώ, ποιες θα είναι οι πολιτικές προϋποθέσεις ε, με τις οποίες θα δεσμεύσουμε, αν θέλετε, αυτή την ε, βοήθεια. Διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δεχτεί ε, άμεσα τις ε, οικονομικές προϋποθέσεις του Δουνουτού. Εμείς όμως θα επιβάλλουμε πολιτικές ε, δεσμεύσεις. Και αυτά τα λέω σε σχέση με αυτά που μας είπατε για τους στρατιωτικούς. Η κυρία Νέτ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Μιγκαρέλη, εδώ είμαι, εδώ είμαι, γιατί δεν άκουσα το πρώτο τμήμα της ε, ομιλίας του, αλλά άκουσα το τέλος όμως. Πρέπει να σας πω ότι και εγώ συμμερίζομαι τις ανησυχίες ε, και τους φόβους των συναδέλφων. Πρέπει νομίζω να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες ή να τις ε, επαναφέρουμε, εάν γίνεται κάτι τέτοιο. Επίσης θα πρέπει να έχουμε κατά νου αυτό το οποίο θα έλεγα το μάθημα από μια πρώτη απόπειρα εκδημοκρατισμού στην Αλγερία πριν από 15 χρόνια περίπου, ότι όταν όλοι οι εξέφρασαν την ανακούφιση τους όταν ακυρώθηκε ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών, διότι στον πρώτο γύρο τα αποτελέσματα δεν μας άρεσαν. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να επαναλάβουμε τώρα. Καταλαβαίνω επίσης και τους συναδέλφους, όπως την κυρία Αναγκόμες που λέει ότι ε, όταν λέμε, πρέπει να πούμε αρκεί κάποια στιγμή, αλλά δεν έχουμε και κανένα συμφέρον να διαλυθεί αυτή η περιοχή. Γι' αυτό πρέπει να σταθμίσουμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση. Έχ, ξέρε, έχετε κάποια γνώμη φαντάζομαι. Μήπως ε, θα μπορούσατε να μας πείτε τι πρέπει να γίνει για να διασφαλίσουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες και τις εκλογικές διαδικασίες. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινήσαμε με την Αραβική Άνοιξη όπου όλοι είμαστε αισιόδοξοι και ε, τώρα μιλάμε για το αραβικό ξύπνημα. Δεν ξέρω τελικά τι από τα δύο θα κρατήσει η ιστορία. Από ό,τι φαίνεται πάντως ε, ο πρόεδρος ε, που θα εκλεγεί από τους ε, αδελφούς μουσουλμάνους ε, έχει μάλλον υποτίθεται ότι έχει εκλεγεί, μπορεί να, να διαλύσει το κοινοβούλιο, τι θα, τι θα, εάν ο πρόεδρος, ο Αιγύπτιος πρόεδρος είναι αυτός θα πάει στο Camp, ε, στο Camp David ε, η, η Βουλή στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, είπε ότι θα αναστείλει τις δημοσιονομικές τη δημοσιονομική βοήθεια. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω τελικά να δούμε τι μπορούμε να στηριχθούμε στον Αιγυπτιακό στρατό ότι θα είναι ουδέτερος και θα, θα προστατεύσει τις πιο ευάλωτες ε, κατηγορίες των πολιτών. Η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή ε, είναι μια οικονομία που έχει γονατίσει. Δεν έχει τουρισμό, δεν έχει βιομηχανία, στηρίζονται στα χρήματα της Σαουδικής Αραβίας. Ε, δεν ξέρω και τι δεσμεύσει ε, ε, ζητάει η Σαουδική Αραβία, τι γίνεται με τους σαλαφιστές. Τέλος πάνω, νομίζω ότι είναι εκρηκτικό το μείγμα. Ευχαριστώ. Ο τελευταίος, ο κύριος Μέιερ. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μιγκαρέλη για τις πληροφορίες που μας έδωσε και ευχαριστώ για αυτό. Χωρίς αμφιβολία περιγράφει μια πραγματικότητα που είναι πραγματικά πολύ απογοητευτική και ισοπεδωτική σε σχέση με την επανάσταση Ταχρήρ και τους στόχους που είχε και τι συνέβη με αυτήν. Και συμφωνώ για, με αυτούς που λένε ότι σε σχέση με την Αίγυπτο έχουμε ένα πραγματικό συνταγματικό πραξικόπημα ενώπιόν μας και το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο και οι Ένωπε δυνάμεις έχουν με διατάγματα προχωρήσει και έχουν ξεπεράσει τα εσκαμμένα και τις αρμοδιότητές τους και αυτά τα οποία έγιναν σε σχέση και με τη διάλυση του σώματος είναι πολύ επιβαρυντικά και σήμερα έχει συγκληθεί και πάλι συνάντηση, διαδήλωση στην πλατεία Ταχρή για να δοθεί απάντηση σε αυτό. Η απάντηση θα πρέπει για να, να επανορθώσει την κατάσταση διότι αν ήταν σε θέση να διώξουν τον ε, Μουμπάρακ γιατί να μην μπορέσουν με τις κοινωνικές δυνάμεις που διαδηλώνουν να προχωρήσουν και να αντιμετωπίσουν αυτό το συνταγματικό πραξικόπημα που είναι παράνομο. Υπάρχει μια φύσα μια πινακίδα στο Ταχρήρ που περιγράφει πολύ καλά την κατάσταση. Λέει, ζητούσαμε ψωμί, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη μας έδωσαν το στρατό, την αστυνομία και τη στρατιωτική αστυνομία. Αντανακλά ακριβώ και τέλεια την πραγματικότητα επιτόπου και θέλουμε οι ίδιοι οι πολίτες οι οποίοι έχουν εξαπατηθεί, εξαπατηθεί σε σχέση με αυτή την τεράστια προσπάθεια που έκαναν να κινητοποιούνται διαρκώς για να διώξουν ένα δικτάτορα. Θα πρέπει να είναι σε θέση αυτή να αντιμετωπίσουν τώρα αυτό το πραγματικό συνταγματικό πραξικό. Μα συμπίπτω μαζί σας και συμφωνώ ότι πραγματικά η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη πραγματικά απογοητευτική και ελπίζω ότι από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε αυτό το συνταγματικό πραξικόπημα να τερματιστεί πλέον. Και κατά κάποιο τρόπο η λαϊκή βούληση, η λαϊκή θέληση να είναι εκείνη η οποία θα πριτανεύσει και θα αναλάβει τα ενία στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ. Ωραία. Ας αφήσουμε τον κύριο Μιγκαρέλη τώρα να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα του κυρίου Σαλαφράκα. Όπως ξέρετε κύριε Σαλαφράκα, ε, κάποιοι εμπειρογνώμονες πήγαν στην Αίγυπτο για να παρατηρήσουν τις εκλογές και να κάνουν συστάσεις με σκοπό τη βελτίωση των επόμενων εκλογών που θα διεξαχθούν. Δηλαδή, αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ε, αποστολή σας στην Αλγερία ή την αποστολή του κυρίου Γκάλε στην Τινησία. Ήταν πολύ λιγότεροι αυτοί οι εμπειρογνώμονες στην Αίγυπτο. Πολύ λιγότεροι. Μια χούφτα άνθρωποι. Αν αυτό σημαίνει ε, με μια χούφτα εμπειρογνώμονες μπορείτε να σχηματίσετε γνώμη. Να απαντήσω, και να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημά σας. Ε, υπήρχαν πολλές οργανώσεις όπως το Carter Center ε, και η αντιπροσωπεία μας επίσης ε, ήταν σε επαφή με όλες αυτές τις οργανώσεις που παρατηρούσαν τις εκλογές Και αυτό που έφτασε τελικά στις Βρυξέλλες ε, από αυτή την εμπειρία ήταν ότι δεν ήταν τέλειες, υπήρχαν ε, περιθώρια βελτίωσης ε, στο επίπεδο της προετοιμασίας των εκλογών και στο επίπεδο της εξαγωγής τους. παρόλα αυτά, παρά τις παρατυπίες, οι παρατυπίες αυτές κατά πάσα πιθανότητα δεν ήταν τόσες και τόσο ισχυρές για να να ανατρέψουν και να ακυρώσουν το αποτέλεσμα. Πρόκειται για εμπειρικά στοιχεία, έτσι, για να μην το πω διαφορετικά. Είχαμε λίγους εμπειρογνώμονες, αλλά χρησιμοποίησαμε το δίκτυο των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των διεθνών οργανισμών που ήταν παρόντες επιτόπου για να δούμε τι πραγματικά συνέβαινε στην Αίγυπτο. Τώρα, αν αμφισβητήσει τα αποτελέσματα των εκλογών ο Σάφικ, τι κάνουμε. Ελπίζουμε όταν η εκλογική επιτροπή θα μιλήσει για τα τελικά, θα πει ποια είναι τα τελικά αποτελέσματα, ο χαμένος να δεχτεί τα αποτελέσματα αυτά. Αν όχι, θα υπάρξει προσφυγή στο συνταγματικό δικαστήριο από τον Τι μπορεί να συμβεί. Υπάρχουν τόσες πολλές υποθέσεις και σενάρια που δεν μπορώ να σας απαντήσω. Θα πρέπει απλούστατα να γίνει σεβαστό το δίκαιο και θα πρέπει οι, οι οι οποίοι προάγουν το δίκαιο να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να εφαρμοστεί η απόφασή τους και να γίνει δεκτή. Εάν δεν γίνει δεκτή, τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχω ιδέα. Πρέπει να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τη δυσκολία την διατύπωσε η κυρία Νέιτ. Ακόμα και αν όλα αυτά δεν μας ικανοποιούν. Ακόμα και αν αηδιάζουμε απέναντι σε αυτή την προδοσία των ιδανικών της Επανάστασης, αν δεν κάνουμε παρόλα αυτά τίποτα και μείνουμε απλοί παρατηρητές μιας οικονομικής επιδείνωσης της χώρας, θα έχουμε πράξει το σωστό, θα έχουμε προάγει τη σωστή πολιτική. Θα... Είναι ένα δίλημα στο οποίο θα βρεθούμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούμε μπροστά σε ένα δίλημα. Θα πρέπει να σταθμίσουμε τα υπέρ και τα κατά της κάθε επιλογής και είμαι σίγουρος ότι η τελική απόφαση δεν θα είναι εύκολη. Τώρα, η ιδανική διαδικασία ποια θα ήταν από την Πέμπτη και μετά να έχουμε ένα πρόεδρο που θα τον δεχτεί ο ιτημένος, ο πρόεδρος αυτός να διορίσει γρήγορα ένα, τον Πρωθυπουργό και την ε, κυβέρνηση, παράλληλα η Συνταγματική Επιτροπή να εκπονήσει το σχέδιο συντάγματος και τους επόμενους μήνες να υιοθετηθεί το σύνταγμα αυτό και να γίνουν ε, Νομοθετικέ εκλογέ, βουλευτικέ δηλαδή εκλογέ. Όλα αυτά είναι εάν αυτό, εάν εκείνο. Αλλά πώ μπορούμε να λειτουργήσουμε και να σκεφτούμε διαφορετικά. Για να περιορίσουμε του κινδύνους μια διολίσθησης, τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι να στρέφουμε συνεχώ το βλέμμα και την προσοχή μα προ την Αίγυπτο και τι αρχέ, να του πούμε ότι σα παρατηρούμε, κοιτάξτε, σα παρατηρούμε. Και κάθε διολίσθηση σε σχέση με τις δημοκρατικές αρχές θα τιμωρηθεί με κάποιο τρόπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά φυσικά ο μοχλός που έχουμε απέναντι σε μια χώρα όπως η Αίγυπτος, ε, ξέρετε, είναι πολύ περιορισμένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς και υπάρχουν πολλοί ε, παράγοντες πολύ πιο σημαντικοί από εμά. Κυρία Γκόμες, ε, το more for more θα πρέπει να οδηγήσει στο less for less. Με ρίσκο θα σας απαντήσω ναι. Αν πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει περισσότερα για χώρες που βρίσκονται σε, αυτή την, που βρίσκονται σε καλή κατάσταση ό,τι αφορά τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, αυτό σημαίνει μηχανιστικά ότι θα πρέπει να μειώσει τη βοήθειά της η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε αυταρχικές χώρες. Αυτό θα συμβεί. Εγώ είμαι γραφειοκράτης. Δεν αποφασίζω εγώ, άλλοι αποφασίζουν. Κυρία Μπραντνερ, μπορούμε να βάλουμε πολιτικές ε, προϋποθέσεις για τη χορήγηση μακροοικονομικής στήριξης. Ξέρετε ότι αυτή η βοήθεια ε, δίνεται σε συμφωνία με το Δούνου του. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι πολιτικοί ηθήνοντες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δώσουν μακροοικονομική στήριξη και βοήθεια σε μια χώρα που στρέφει την πλάτη στη δημοκρατική μετάβαση. Μπορεί να κάνω λάθος με αυτό που λέω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Προφανώ δεν είναι τεχνική η απόφαση. Καταρχά θα πρέπει να ληφθεί μια πολιτική απόφαση, να γίνει μια πολιτική αποτίμηση τη ε, διαδικασία τη μετάβαση και μετά θα ληφθεί η τεχνική απόφαση να δοθεί, να χορηγηθεί αυτή η μακροοικονομική βοήθεια. Μην ξεχνάτε επίση ότι αυτή την απόφαση δεν την παίρνουν οι γραφειοκράτε. το Συμβούλιο αποφασίζει και εσείς έχετε, εσείς ως Ευρωκοινοβούλιο συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα υπάρξει αυτή η πολιτική εκτίμηση τη στιγμή που θα αποφασίσουμε, που θα δούμε πρέπει να δώσουμε αυτή την ε, μακροοικονομική βοήθεια ή όχι. Και πάλι, ενέχε, ε, υπάρχει ο κίνδυνος να κάνω λάθος. Αλλά δεν νομίζω. Ε, κυρία Νέη, τι μπορούμε να κάνουμε για να διατηρήσουμε την εκλογική διαδικασία, συνεχής επαφή με όλους και με τους στρατιωτικούς και να τους πούμε ότι αν προδώσουν τα ιδεώδη της Επανάστασης, σκάφουν το λάκκο τους. Γιατί χρειάζονται κάποιου εξωτερικούς εταίρους και συμμάχους και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από αυτούς. Και μέσα από το διάλογο και την πειθό μπορούμε να ελπίζουμε, ελπίζω, ελπίζουμε και το τονίζω το ελπίζουμε, ότι μπορεί να επηρεάσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα επιτρέψουν την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας η στρατιωτική. Κύριε Τάνοκ, για το Camp David. Επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά στους ε, Αιγύπτιους ομόλογους μας ότι πρέπει να, δεσμευτούν, να σεβαστούν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις. πρώτη από αυτές είναι να ε, σεβαστούν την ε, ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ. Θα μου πείτε δεν είναι αρκετό. Είναι απλώς μια αρχή. Και σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις συναντήσεις, μιλάμε για αυτές τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει οι Αιγυπτοί. Και ότι δεν θα ήταν προς το συμφέρον κανενός η Αίγυπτος να ξεχάσει, να ακυρώσει, να στρέψει την πλάτη σε αυτές τις διεθνείς υποχρεώσεις, λόγω της βιοστρατηγικής της σημασίας. Κατ' εξαίρεση. Κατ' εξαίρεση μπορούμε να δεχτούμε και άλλες ερωτήσεις. Δεν νομίζω ότι ζητάει κανείς άλλο το λόγο. Περνάμε στο επόμενο σημείο, όμως καταρχάς να σας πω ότι η, η αποστολή του Μπαχρέιν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας είπε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Μπαχρέιν ε, ανέβαλε την επίσκεψή του διότι θα πρέπει ε, να συμμετέχει η χώρα του στο πένθος λόγω του θανάτου του Σαουδάραβα πρίγκιπα. Το σημειώνουμε αυτό και περνάμε στο επόμενο σημείο. Ε, τώρα να σας ενημερώσω ότι τα αραβικά μπορεί να ακουστούν από την καμπίνα νούμερο 17. 17. Πάμε στο επόμενο σημείο που αφορά την ανταλλαγή απόψεων με, για την Συρία. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να ε, ε, καλωσορίσω τους τρεις ε, ομιλητές μας, συγητές μας. Η κυρία Αμαλάχ θα έρχεται, ο κύριος Καμάλα Λαλμπουάνη, κάθε δίπλα μου, ε, μέλος της Συριακής Αντιπολίτευσης έχει συλληφθεί, έχει κρατηθεί από το 2005 2011 από τις, ε, το καθεστώς ε, του Ελάσαντ είναι ιδρυτής του Πατριωτικού Μετόπου που είναι μια συνιστόσα της Συριακής Αντιπολίτευσης και ο κύριος ο Σαμ Αλκατράμπη είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Συρίας και η κυρία Αϊτά Μαλμαλάχα, την οποία θα δούμε σε λίγο, είναι μέλος της αντιπολίτευσης, έχει συλλευθεί την δεκαετία του, το 2010 του του 80, συγγνώμη, από, την, ε, από το καθεστώς Άσαντα Ε, επίσης, ε, να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Μιγκαρέλη, ο οποίος θα μας βοηθήσει ε, σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων και θα μας μιλήσει και για τον Παχραήν αργότερα. Και να ξεκινήσω λέγοντας ότι η κατάσταση στην Συρία είναι τραγική. Η βία έχει εξαπλωθεί παρά τις προσπάθειες παρέμβασης από την ε, διεθνή κοινότητα. Έχουμε φτάσει σε έναν εμφύλιο πόλεμο. Έχουν, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, κάνει πολύ πιο αυστηρές τις κυρώσεις προς το καθεστώς. Οι κυρώσεις όμως αυτές φαίνεται ότι δεν έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην, στο καθεστώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε να παρέμβει πιο έντονα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά μέχρι στιγμής ήταν αδύνατο να πείσουμε την Ρωσία δράτω με της ευκαιρίας ε, για αυτή την, από αυτή την ανταλλαγή απόψε να καταλάβω. Θα σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηρίξει πιο αποτελεσματικά την ε, ανέβρεση μιας ε, ειρηνικής λύσης στα προβλήματα της Συρίας. Πόσο κοστίζουν, αν θέλετε, τα συμφέροντα, της, ε, τα πολιτικά και θεωρητικά συμφέροντα της Ρωσίας ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση και μιλάω και για το ναύσταθμο. Ε, ποιες είναι οι στόχοι της αντιπολίτευσης και ποιες είναι οι δυνατότητες όλα αυτά, όλες αυτές οι συνιστώσεις της αντιπολίτευσης να δημιουργήσουν μια ενιαία ομάδα και ποια είναι η, ποιο είναι το βάρος της ε, θρησκευτικής συνιστώσας αυτή τη στιγμή και ποια, πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί για το μέλλον της, το μέλλον της Συρίας. Και θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους συζητητές να μην ξεπεράσουν τα πέντε λεπτά. Ήρθε ο κύριος Άιτα Μαλμαλάχα, το ήθελα να τον καλωσορίσω. E eh, inizio eh, con lei. Cinque minuti per... Λοιπόν, πέντε λεπτά έχει ο καθένας για την παρέμβασή του. Σούκρα. Thank you so much. This is the second time I have been... Είναι η δεύτερη φορά που είμαι εδώ, αυτό το μήνα. Ήμουνα εδώ το 2005 με τον κύριο Μπράντα και άλλους ήμουν σε σχέση με την Προεδρία επί μεγάλο χρονικό διάστημα είμαστε υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας των πολιτών στη Συρία. Αυτά που συμβαίνουν στη Συρία δεν είναι μόνο μια εκδηλή κρίση που πρέπει να σταματήσει το δυνατόν ταχύτερα και με οποιαδήποτε μέσα είναι πραγματικά υπόθεση ανθρωπιστικής ασφάλειας αλλά και επίσης είναι μια πραγματική επανάσταση. Επανάσταση που προσπαθεί να ανοίξει πόρτες και πύλες στην αλλαγή, στην ανατροπή, απόλυτη αλλαγή και ανατροπή του καθεστώτος και της πολιτικής ζωής, αλλά και του πολιτισμού στην Συρία. Η κοινωνία των πολιτών και οι πολίτες της Συρίας θέλουν να δημιουργήσουν μια νέα προοπτική ιστορική για την περιοχή μας. Η Μέση Ανατολή τώρα αποτελεί το άθροισμα και τη σύνοψη ενός προβλήματος που έχει εκραγεί παγκόσμια και αυτά τα οποία θα συμβούν εκεί θα έχουν επιπτώσεις παγκόσμιες. Γι' αυτό πρέπει η δημοκρατία και η ελευθερία να επιβληθούν στη Συρία και σας καλούμε να υποστηρίξετε τους Σύριους να επιτύχουν την ελευθερία τους και την απελευθέρωσή τους. Θα δείτε τότε, θα βρείτε ότι έχετε φίλους στη Συρία. Υπάρχουν σενάρια διαφορετικά. Πρώτον, να υπάρχουν, να, είναι κατακαιρματισμένοι οι Σύριοι και να πολεμούν ο ένας τον άλλον και το άλλο σενάριο να ενωθούν και να απελευθερωθούν. Πρέπει να βοηθηθούν οι Σύριοι να δημιουργήσουν τη νέα μελλοντική τους προοπτική ως σενάριο και να συνεργαστούν με άλλα κράτη στο πνεύμα του πολιτισμού και της ειρήνης που πρέπει να πριτανεύσουν. Στη σημερινή κατάσταση πρέπει να δεχθούμε ότι οι Σύριοι έχουν το δικαίωμα να αυτοϊπερασπίζονται, να αυτοϊπερασπιστούν και να αμυνθούν και πρέπει να τους βοηθήσουμε να το κάνουν. Να, το κάνουν. να πιστεύουν ότι έχουν το δικαίωμα αυτό, πώς μπορούμε να τους αρνηθούμε το δικαίωμα να αυτοαμυνθούν και να αυτοπροστατευτούν και πώς μπορούμε να μην τους ε, βοηθήσουμε να προστατευτούν από τις ομότητες του παράνομου αυτού καθεστώτος ε, που έχει και εξωτερική υποστήριξη. Πρέπει να επιβληθεί η δικαιοσύνη. Αν όμως αρνηθούμε αυτή την προοπτική αρνηθείτε εσείς στη Συρία αυτή την προοπτική θα πρέπει να συνεχίσουμε να αμυνόμαστε. Γιατί όποιο και να είναι το αντίτιμο ποτέ δεν πρόκειται να ξαναδεχθούμε ένα δικτατορικό καθεστώ και να ζήσουμε υποδικτατορία Δεν είναι μια κατάσταση λοιπόν όπου μπορεί να δοθεί γρήγορα μια λύση. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε σταθερότητα και ειρήνη με άλλο τρόπο, με ένα άλμα εκτός αν υπάρχει το θάρρος από πλευρά σας να μας βοηθήσετε να κατακτήσουμε τη δημοκρατία και την πολιτισμική πολιτιστική μεταρρύθμιση. Μια νέα δημοκρατική Συρία όπως ζητούμε πρέπει να σέβεται όλες τις ομολογίες και τις θρησκείες και σε ένα πλαίσιο ασφάλειας. Δεν είναι το Ιράκ, η Αιγύπτος, η άλλη χώρα ή η Συρία. Μπορεί να συνενωθούν όλες οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, αλλά ακόμα αυτό δεν έχει επιτευχθεί. Χρειαζόμαστε οποιαδήποτε δυνατότητα ειρηνικής επίλυσης, αλλά πρώτη προϋπόθεση και κύρια προϋπόθεση είναι η δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος χωρίς αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Χρειαζόμαστε βοήθεια από τους φίλους και τους γείτονές μας. Υποστήριξη από όλους, όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο από ένα κόμμα ή ομάδα. Χρειαζόμαστε βοήθεια για να προωθηθεί και προαχθεί η δημοκρατία και να μην κρατηθεί και ανανεωθεί η δικτατορία. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Αλμαλάχ, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την πρώτη φορά ε, μιλήσαμε μέσω του Skype. Πέρυσι ήρθα φυσικός πώς ε, για μια συνάντηση εδώ και σήμερα είναι η τρίτη φορά που έρχομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρετε ότι τι συνέβη στη Συρία μέχρι τώρα, σφαγές παντού. Η καταστολή που υπάρχει σε όλες τις ε, πόλεις, σε όλες τις κομμουπόλεις, σε όλα τα χωριά. Έχουμε απέναντί μας τη Διεθνή Επιτροπή, η οποία όμως δεν έκανε τίποτα για να υποστηρίξει τη Συρία. Λόγω του βέτο της Ρωσίας. Υπάρχει συνεργασία με τη Ρωσία, το Λίβανο, ε, το Χεσμολά στο Λίβανο και τη Συρία και μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί πάνω από 20.000 άτομα. 250.000 είναι στις φυλακές και 1,5 εκατομμύριο είναι πρόσφυγες. Επομένως, όποιος κάνει λόγο για διαπραγματεύσεις και για διάλογο με το καθεστώς, πλανάτε πλάνη Είναι αδύνατο κάτι τέτοιο. Ίσως η Ρωσία πιστεύει ότι το καθεστώς του Μπασάρ είναι παρελθόν. Ίσως το πιστεύει. και το Ιράν όμως. Και ο Υπουργός Εξωτερικών θέλησε, του Ιράν, θέλησε να με συναντήσει. Εγώ αρνήθηκα να πάω και στο Ιράν και στη Ρωσία. Τώρα, στη Συρία δεν υπάρχει καμία πολιτική προοπτική λόγω της συνεργασίας της Συρίας και του Ιράν. Α, συγγνώμη, πέρασα στα αραβικά, χωρίς να το καταλάβω. Πέρασα στη μητρική μου έτσι. Σκεφτόμουν αραβικά και μίλησα αραβικά. Μπορείτε να μιλήσετε αραβικά. Ε, τότε να, συμφωνεί, να συνεχίσω στα αραβικά. Έλεγα λοιπόν ότι η διεθνής ε, κοινότητα ε, κοιτάζει την ε, Συρία και τον Συριακό λαό ως μια διαιρεμένη κοινωνία. Να θέσω το παρακάτω ερώτημα. Ξέρετε μια χώρα, ένα λαό στον κόσμο όπου όλοι σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, όπου υπάρχει απόλυτη ενότητα στο λαό. Εμείς στη Συριακή Αντιπολίτευση δεν έχουμε όλοι τις ίδιες απόψεις ίσως, αλλά συμφωνούμε επί κάποιων βασικών και θεμελιωδών αρχών. Δηλαδή θέλουμε ένα δημοκρατικό καθεστώς πάνω απ' όλα στη Συρία. Θέλουμε νομοθετικές εξουσίες. Θέλουμε δικαστικές εξουσίες ανεξάρτητες. Φυσικά στην Συριακή Αντιπολίτευση υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις σε ό,τι αφορά το ρόλο του στρατού σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, αλλά παρά τις διαφορές αυτές συμφωνούμε επί κάποιων θεμελιωδών αρχών. Όπως ξέρετε, πρόσφατα συναντηθήκαμε στην Κωνσταντινούπολη και δημιουργήσαμε μια επιτροπή από πολλές προσωπικότητες Συρίων, ε, αντιπολιτευόμενους, ούτως ώστε να ετοιμάσουμε μια μεγάλη ε, διάσκεψη ε, που θα λάβει χώρα στο Κάιρο, στην Αίγυπτο προκειμένου να, λάβουμε, ε, να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα για να υπάρξει μια ενότητα στην αντιπολίτευση. Και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Δεν θα υπάρχει κανένας λόγος πια η διεθνής κοινότητα να μην μας δώσει τη βοήθεια που ζητάμε. Μετά από 15 ολόκληρους μήνες σφαγών, φρικαλαιοτήτων, πάσης φύσεως. Θέλω να επανέλθω σε αυτά που είπε ο κ. Καμάλι Στη Συρία Υπάρχουν πολλές δοξασίες θρησκευτικέ. Υπάρχουν όμως κυρίως ε, θρησκευτικές Αλλά δεν υπάρχει όμως ε, μία, ένας ιστός, ας πούμε, ε, μεταξύ, και μία ενότητα μεταξύ αυτών. Να σας πω, επί παραδείγματι, ότι ένας παλιός υπουργός της Συρίας, που ήταν χριστιανός, και επί πολλά χρόνια ήταν πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου. Επίσης υπήρχε και ένας υπουργός θρησκευμάτων από άλλο θρησκευμά. Δεν ήταν χριστιανός. Ε, τα προβλήματα που γνωρίζουμε σήμερα, που βλέπετε σήμερα, τα δημιούργησε το καθεστώς, όχι οι διάφορες ε, κοινότητες, όχι οι διάφορες θρησκευτικές μειονότητες. Πρέπει να σας πω ότι ο Συριακός λαός είναι μοναδικός στις φιλοδοξίες του, στα αιτήματά του για μεγαλύτερη ελευθερία. Τι εννοώ. Θέλω να σας πω ότι ο λαός μας δεν είναι ένας λαός που βασίζεται στις θρησκευτικέ πεπιθήσεις. Δεν βασιζόμαστε στις θρησκευτικέ δοξασίες και δεν, δεν είναι χτισμένη έτσι η κοινωνία μας. Φυσικά, ορισμένοι διεθνείς φορείς μιλάνε για το θρησκευτικό χαρακτήρα της χώρας και τις θρησκευτικέ μας πεπιθήσεις. Όταν έγιναν διαπραγματεύσεις μεταξύ της Γαλλίας και των Συρίων στο παρελθόν, οι Σύριοι είχα ζητήσει όταν ολοκληρωθεί η γαλλική εντολή, κανένας να μην ε, διωχθεί λόγω της θρησκείας του. Κανένας Σύριος. Αυτό έχει γίνει στο παρελθόν ε, της Συρίας. Αυτή είναι η ιστορία μας. Η κυρία Αλκατράμπη. Ο κύριος, συγγνώμη. Καλημέρα. Θα ήθελα να χαιρετήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Να σας ευχαριστήσω γιατί μας επιτρέψατε να έρθουμε εδώ. Ε, είναι η πρώτη φορά που απευθύνομαι την, ε, σε μέλη του Κοινοβουλίου. Εδώ και δεκαετίες, ε, τέσσερις δεκαετίες ε, το καθεστώς μας, το καθεστώς στην Συρία ήταν, περνούσε από τον πατέρα στο γιο και επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω τι συνέβη τους τελευταίους 15 μήνες. Ο λαός της Συρίας αποφάσισε επευκαιρία του, της Αραβικής Άνοιξης ε, να, να πάρει στα χέρια του το μέλλον του. Δεν ε, γνωρίσαμε ποτέ την ελευθερία. Καμιά μορφή ελευθερίας. Το καθεστώς πολλές φορές ε, απέδειξε ότι δεν θέλει ανοίγματα προς εξωτερικό. Απαγόρευσε τις αποστολές των ΗΕ, δεν δέχτηκε την αποστολή της ε, Αραβικής Λίγκας, ε, δεν τους επέτρεψαν να, καλύψουν, να δούνε τις προβληματικές περιοχές, δεν επέτρεψε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να καλύψουν τα επεισόδια ούτε την Αραβική Λίγκα, ούτε την, τον Αραβικό Σύνδεσμο, συγγνώμη, ούτε την, το, τον ΟΗΕ, ε, στον ΟΗΕ επέτρεψε να επισκεφθούν τις περιοχές και να δει ο κόσμος τι ακριβώς ε, συμβαίνει. Τώρα αναστέλλεται η αποστολή των παρατηρητών των ΗΕ. Αυτό το οποίο διαπράττει το Συριακό καθεστώς είναι η σφαγή του πληθυσμού και η σφαγή αυτή αποδεικνύει σε όλο τον κόσμο ότι το καθεστώς αυτό δεν ενδιαφέρεται για, το, για τους πολίτες της χώρας. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να κρατήσουν την εξουσία με κάθε τρόπο. Το καθεστώς έχει δείξει το πρόσωπό του, έχει δείξει τι μπορεί να κάνει. Έχουμε ε, φυλακίσεις ε, αυθαίρετες, ε, έχουμε σφαγές, έχουμε βασανιστήρια και όλα αυτά τα γεγονότα θα πρέπει να τα συνδυάσουμε και με τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό των στρατιωτικών που έρχονται στον ελεύθερο Συριακό στρατό. Θα πρέπει δηλαδή να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατευτούμε από αυτό το καθεστώς και από τις αυθαιρεσίες του. Το καθεστώς προσπάθησε με διάφορους τρόπους να δείξει ότι θέλει κάποια ανοίγματα. Επελευθέρωσε, απελευθέρωσε κάποιους φυλακισμένους, αλλά όχι όλους και στην αποστολή του Κόφι Ανάνα και στις, στο πρόγραμμα του Κόφι, στην πρόταση του Κόφη Ανάνα ε, προσπάθησαν να απαντήσουν ε, απελευθερώνοντας κάποιους, όχι όμως όλους και ακόμα ε, έχουμε πολλούς φυλακισμένους. Το καθεστώς έχει τρομοκρατήσει τους πολίτες, έχει τρομοκρατήσει το λαό και ε, αυτό το οποίο προσπαθεί να δείξει τώρα είναι ότι οι πολίτες δεν θέλουν την ελευθερία, δεν θέλουν την, ε, τον, δημοκρατία, θέλουν το χάος. Ε, όμως αυτό το οποίο ουσιαστικά συμβαίνει είναι ότι το καθεστώς θέλει καμένη γη η στάση της Ρωσίας με το βέτο του Συμβούλιο Ασφαλείας δεν βοηθάει το λαό της Συρίας. Η διατήρηση του σημερινού καθεστώτος ε, θα μπορούσε να, μάλλον το καθεστώς αν θέλετε, θα μπορούσε να, να το παρομοιάσουμε με τους Ναζί ή με το καθεστώς του Μιλόσεβιτς πιο πρόσφατα κτλ. Ε, εδώ και 40 χρόνια βρίσκεται στην εξουσία το καθεστώς αυτό και έχει κάνει πολλές σφαγές. Έχει στο παρελθόν ε, ε, διαπράξει εκατοντάδες σφαγές, έχει φυλακίσει κόσμο και αυτό το οποίο εμείς ζητάμε είναι, την, η ελευθερία μας. Θέλουμε μια ειρηνική λύση στα προβλήματα της Συρίας. Επιζητούμε μια ειρηνική λύση, επαναλαμβάνω, διότι θέλουμε ο λαός μας να πάρει την ε, μοίρα του στα χέρια του. Ευχαριστώ. Ωραία. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους, ο κύριος Μιγκαρέλη θα μας ε, πει τις απόψεις του και θα μας ε, ενημερώσει για την, τις απόψεις Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λίγα λεπτά μόνο να σας ενημερώσω ε, γιατί όπως και εσείς τώρα μάθαμε ότι ο στρατηγός ο οποίος ε, ε, ηγείται της αποστολής ε, των, των Ηνωμένων Εθνών ανέστηλε τις δραστηριότητες της αποστολής λόγω ακριβώς της αναζωγόνησης αν θέλετε των ανθρωπραξιών και αυτή η αναζωγόνηση είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχήσει διότι φαίνεται ότι ελοχεύει ο κίνδυνος ενός εμφυλίου πολέμου όπως επίσης και ένας ε, και ο κίνδυνος θρησκευτικού πολέμου, διότι ήθελε να βάλει και μια θρησκευτική πτυχή, αν θέλετε, ο Ασάντ στα όλα αυτά τα θέματα. Ε, και μάλλον θα το πετύχει. Όλα αυτά, επομένως, είναι ανησυχητικά και για τη Συρία, αλλά και για όλη την περιοχή. Ξέρουμε ότι το σχέδιο του Κόφη Ανάνα δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί πλήρως. Παρόλα αυτά, όμως, είναι η λιγότερο κακή προπτυχή η βρίσκεται αυτή τη στιγμή τα πάνω στο τραπέζι αν θέλουμε να έχουμε μια πολιτική λύση. Γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει και συνεχίζει να υποστηρίζει το σχέδιο του Κόφι Ανάν. Όπως επίσης ε, χαιρετίζουμε και την πρωτοβουλία ε, η παρουσία να δημιουργήσουν μια ομάδα ε, επαφής η οποία θα συνεδριάσει 30 Ιουνίου στην Γενέβη και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι θα πρέπει να έχουν ένα συνεχή διάλογο με τους ε, Δυτικούς για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια κοινή άποψη, μια κοινή δράση έτσι ώστε να καμφθεί το καθεστώς Ασάντα. Λοιπόν, ε, από όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ζητάμε να λάβουν ε, υπόψη όλα τα στοιχεία για να υποστηρίξουν το σχέδιο ΑΝΑΜ και κυρίως εν ώψη της 19 η Ιουλίου ε, όπου θα συζητηθεί ε, όπου θα συζητηθεί η διεύρυνση του, της αποστολής των παρατηρητών. πρέπει τα Ηνωμένα Έθνη να αποφασίσουν τι θα κάνουν ε, για αυτή την, με αυτή την αποστολή. Επίσης ε, θα πρέπει να γίνει πιο στενό, πιο έντονος, πιο, πιο δραστήριος αν θέλετε και ενεργός ο διάλογος με την Ρωσία και την Κίνα ε, γιατί αυτές οι χώρες μπορούν να αντιστρέψουν τις, τις εξελίξεις, μπορούν να ανατρέψουν μάλλον τα, την κατάσταση και να γύρει η πλάστικα από τη μια ή από την άλλη πλευρά. Τώρα, όσον αφορά την αντιπολίτευση, αυτό το οποίο σας ζητάμε κύριοι δεν είναι να ενωθείτε, ξέρουμε ότι έχετε διαφορές και είναι σωστό αυτό. Όμως αυτό το οποίο θέλουμε είναι να μπορέσετε να δημιουργήσετε μια κοινή πλατφόρμα για τον καλύτερο τρόπο να, ε, για να έχουμε ένα, καλύτερο, ένα καλό τρόπο να προωθήσουμε τις μια πολιτική λύση. Διότι αν δεν υπάρχει μια ελάχιστη ε, απόφαση για τις πολιτικές εξελίξεις τότε η, αυτή η μετάβαση ε, σε ένα δημοκρατικό καθεστώς δεν θα μπορέσει να γίνει. Επομένως δεν σας ζητάμε να δημιουργήσετε ένα κίνημα, ένα κόμμα γιατί αντιπροσωπεύετε πολιτικές απόψεις, εθνικές απόψεις, εθνική, έχετε εθνική προέλευση διαφορετική, ανήκετε σε διαφορετικές θρησκείες, άρα δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κίνημα. Όμως όταν θέλετε να δώσετε μία μάχη σε ένα αυταρχικό καθεστώς πρέπει να έχετε ένα κοινό όραμα ε, όσον αφορά το την μετάβαση και το μεταβατικό στάδιο και το που θέλουμε να πάμε. Κάτι το οποίο έκαναν στην Λιβύη, τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αρκούν αυτά που κάνουμε, παρόλα αυτά ε, υποστηρίζουμε την αποστολή, έχουμε... 8 εκατομμύρια, έχουμε δεσμεύσει 8 εκατομμύρια για 25 άρματα. Ε, επίσης ε, υποστηρίζουμε και, και κάποιες άλλες ε, δραστηριότητες επιτόπου. Ε, επίσης δεσμεύουμε κονδύλια για να ενισχύσουμε τον διάλογο ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκομένους. Όσον αφορά την ανθρωπιστική πτυχή, θέλουμε να, η συμφωνία ανάμεσα στον ΟΗΕ και την Συρία, έτσι ώστε να καλυφθεί το 1 εκατομμύριο άτομα να υιοθετηθεί. Έχουμε 32 εκατομμύρια ευρώ 10 εκατομμύρια από την ΕΚΟ και 20 εκατομμύρια από τα κράτη-μέλη που έχουμε συγκεντρώσει. Δεν είναι πολλά τα χρήματα, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα σημαντικό ποσό. Επίσης αποφασίσαμε να αυξήσουμε την βοήθεια προς τις οργανώσεις ε, προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία ε, ε, Εγκρίναμε ένα κονδύλι 23 εκατομμυρίων ευρώ για τους πρόσφυγες που, του Σύριους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις γειτονικές χώρες. Επίσης, η Υπουργείο των Εξωτερικών που θα συνεδριάσουν την επόμενη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο, για άλλη μια φορά ε, θα αναφερθούν στην, ε, στις στο, στο γεγονός ότι θα πρέπει οι κυρώσεις να γίνουν πιο αυστηρές, αλλά με ένα τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να θίξουν την κυβέρνηση και όχι τον λαό της Συρίας. Ευχαριστώ κύριε Μιγκαρέλη. Ε, πολλοί ζητούν το λόγο. Ε, θα έχουμε δύο ομίλους ομιλητών. Ο κύριος Σαλαφράγκα είναι ο πρώτος από τον πρώτο όμιλο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να καλωσορίσω και να χαιρετήσω την παρουσία των προσκεκλημένων μας εδώ. Όπως είχαμε ήδη ευκαιρία να συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε στο Στρασβούργο με την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, τα όσα είπαν για να χαρακτηρίσουν την κατάσταση στην Συρία είναι ανυμπόρια, απόγνωση, απογοήτευση. Γιατί να μην το πούμε, ανυμπόρια, αδυναμία της διεθνούς κοινότητας να αντιμετωπίσει και να αναχαιτήσει αυτή τη βία τις βιοπραγίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Πρόεδρος πολύ καλά επεξήγησε στην εισαγωγή του τις προσπάθειες που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για να πετύχει εναλλακτική υιοθέτηση, υιοθέτηση εναλλακτικών μέτρων. Το σχέδιο του <clears throat> Κόφι Ανάν ήταν θνησιγενές. Πέθανε προτού καν μπορέσει να αναπτυχθεί. Και σε σχέση με τα όσα αναφέρθηκαν ο κύριος Ασάντ, πρόεδρος Ασάντ, θέλησε να κερδίσει χρόνο με αυτό για να συνεχίσει διαρκώς να αυξάνει τον αριθμό των θυμάτων με τις βιοπραγίες του. Η ερώτηση που διατύπωσε ο πρόεδρος στην αρχή της συνεδρίασης είναι απόλυτα σχετική και σημαντική. Τι μπορεί να κάνει η διεθνή κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεδομένου του βέτο της αρνησικυρίας της Ρωσίας και της Κίνας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για να τερματιστεί αυτή η κατάσταση στη Συρία. Εγώ πιστεύω πέρα από απαιτήσει όσον αφορά την αντιπολίτευση ή τους αντιφρονούντες, οι απαιτήσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι σαφείς και κάθετες στους ίδιους τους υπεύθυνους αυτής της κατάστασης, που είναι το καθεστώς Ασάντ. Σε αυτό το πλαίσιο μια ερώτηση, Πρόεδρε, που θα ήθελα να διατυπώσω προς τους προσκεκλημένους μας. Η ερώτηση είναι, αυτός ο πολλαπλασιασμός ομάδων επαφών που παρατηρείται, είναι μια λύση, βιώσιμη λύση. Και χωρίς την παρουσία σε αυτή την ομάδα επαφών όπως πρότεινε η Ρωσία του Ιράν, είναι σκόπιμο να γίνεται κάτι τέτοιο ή όχι. Οι Ηνωμένε Πολιτείε προφανώ το απορρίπτουν αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να γνωρίζω εσεί τι πιστεύετε. Πιστεύετε ότι κάποιε πρωτοβουλίε όπω η πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών τη Γαλλία, τη ε, προηγούμενη κυβέρνηση ή του νέου Υπουργού Εξωτερικών τη Γαλλία θα μπορούσαν να είναι σοβαρέ εναλλακτικέ βιώσιμε λύσει για να σταματήσει αυτή η φοβερή, τρομερή κατάσταση στη Συρία που όπω αναφέρθηκε δείχνει την απογοήτευση την απόγνωση, την οργή και την αδυναμία της διεθνούς κοινότητας για να εξευρεθεί κάποια λύση που δεν μπορεί να βρεθεί για να τερματιστεί αυτή η κατάσταση εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράνκα και σας ευχαριστώ που σεβαστήκατε τόσο ωραία τον ε, χρόνο που σας έδωσα. Κυρία Γκόμες για τρία λεπτά. Έχω, αισθάνομαι απόλυτη αλληλεγγύη με το Συριακό λαό. Και αυτό σημαίνει ότι καταρχήν θεωρούμε ότι έχει το δικαίωμα ο Συριακός λαός να υπερασπίσει τον εαυτό του. Υποστηρίζουμε ότι το καθεστώς του Ασάντ και ο ίδιος ο Ασάντ, αν επιβιώσουν, θα πρέπει να προσαχθούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για αδικήματα πολέμου, αδικήματα κάτω ανθρωπότητας. Και βέβαια, η διεθνής κοινότητα έχει το... την υποχρέωση να σας υπερασπιστεί, αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο γιατί η Ρωσία βλοκάρει το Συμβούλιο Ασφαλείας και η Κίνα, αλλά κυρίως η Ρωσία είναι υπεύθυνη. Παρ' όλα αυτά, η διεθνής κοινότητα θα μπορούσε να κάνει κάτι, να κάνει αυτά που δεν έκανε στη Ρουάντα, ενώ έκανε κάποια πράγματα για το κοσφοπέδιο. Δυστυχώς. Και ας μην μιλάμε και επανερχόμαστε ξανά και ξανά σε αυτό το περιβόητο σχέδιο ΑΝΑΝ, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι του ΑΝΑΝ λένε ότι το σχέδιο αυτό είναι αναποτελεσματικό. Δυστυχώς υπάρχει μια πλειάδα παραγόντων αρνητική για όλους μας, όχι μόνο για τους Σύριους που πληρώνουν και το τίμημα. Η, τραγεδ... η τραγωδία για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι ε, είμαστε σε περίοδο κρίσης και άρα εμφαλοσκοπούμε. Οι Αμερικανοί έχουν τις εκλογές τους, ε, οι γείτονε της ε, Συρίας, το Ιράν κτλ. προτιμούν το διάβολο που ξέρουν τον Ασάντ για διάφορους λόγους. Η τραγωδία είναι ότι είναι εντελώς ανίσχυρη η ανίσχυρος ο Αραβικός Σύνδεσμος, μην ξεχνάμε και ότι τον εμποδίζει και η Ρωσία. Και τώρα μπαίνω στην Αίγυπτο τη Συρία. Έχετε και εσείς κάποια εσωτερικά εμπόδια, είσαστε τόσο κατακαιρματισμένοι η αντιπολίτευση. Στη Λιβύη, όπως είπε ένας ομιλητής, ήταν πολύ αποφασιστικό το γεγονός ότι ενώθηκαν με σκοπό να ξεφορτωθούν τον δικτάτορα. Ένα εθνικό σκοπό. Εσείς, αγαπητοί φίλοι, τι μπορείτε να κάνετε για να δημιουργήσετε αυτή την ενότητα στην ε, αντιπολίτευση, ούτω ώστε να είσαστε κι εσεί τόσο αποτελεσματικοί για να διώξετε το καθεστώ και να επιλύσετε τι διαφορέ σα μετά, ε, ούτω ώστε να μπείτε σε μια δημοκρατική διαδικασία. Ευχαριστώ. Mr. Uh, President... Uh, Ευχαριστώ. Πρόεδρε, λέει η κυρία Νέιτς. Θέλω να καλωσορίσω τους τρεις Σύριους φίλους μας Ορισμένοι δεν είναι εδώ για πρώτη φορά. Σας γνέφω που είμαι, εδώ στο μέσο της αίθουσας. Δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέφθησε το σώμα αυτό. Εκ μέρους τη πολιτικής, μου ομάδα θα ήθελα επίση να σα εκφράσω και εγώ την αλληλεγγύη μου, προσωπική και πολιτική της ομάδας μου, ε, ως προς τον αγώνα σας, Δεν θέλω να μακρηγορήσω για να παρουσιάσω την απογοήτευση, την αδυναμία που αισθανόμαστε ε, για το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να κάνει τίποτα αυτή τη στιγμή λόγω της αρνητικής στάσης της Ρωσίας και της Κίνας Συμβούλου Ασφαλείας στο ΙΑ. Αλλά για να μιλήσω τώρα πιο ομά. Νομίζω ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε βέτο από τη Ρωσία και την Κίνα, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε όρεξη για στρατιωτική επίθεση στη Συρία, για εισβολή στη Συρία. Να σας θέσω μια ομή ερώτηση. Ο κύριος Λαγκουάμι ε, ζήτησε να εξευρεθεί μια ειρηνική λύση. Πώς τη βλέπετε. Φυσικά οι Σύριοι έχουν το δικαίωμα να πάρουν τα όπλα και να προστατευτούν. Αλλά για μας το δίλημα είναι εξωτερική παρέμβαση ναι ή όχι. Μακάρι να μην ήταν απαραίτητη και να μην είναι απαραίτητη. Αυτό είναι το ιδανικό για μας. Εσείς πέστε μας πώς το βλέπετε, πώς αισθάνεστε, πώς βλέπετε αυτό το δίλημα που νομίζω ότι το έχετε κι εσείς, αλλά το βλέπετε από την πλευρά σας. Τέλος. Εκ μέρους της ομάδας μου θέλω να υποστηρίξω τις εκκλήσεις που γίνονται. Όχι να ενωθείτε εσείς ε, σε ένα ενίο κίνημα της αντιπολίτευσης, γιατί αυτό είναι μη ρεαλιστικό, δεν είναι καν δημοκρατικό. Να έχετε όμως μια ελάχιστη πλατφόρμα για να ξέρετε που θέλετε να πάτε και για το πώς θα πάτε εκεί που θέλετε να πάτε. Αυτό ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για σας. Κυρία Μπράτνερ. Ευχαριστώ. Κύριε Μιγκαρέλη, φέρατε κάτι. Είναι η 17η φορά που επιβάλλουμε κυρώσεις. Εδώ υπάρχουν και θέματα κονδυλίων. Είναι κρίμα που κάνουμε τόσο λίγα πράγματα για τη Συρία. Αν τον περασμένο Ιούνιο είχαμε ένα κατάλογο με 200 άτομα που θα τους επιβάλαμε κυρώσεις, αν είχαμε πάρει αυτή την απόφαση, δεν μιλάω για να κυρώσουμε κάποιον γιατί επιχειρηματία, πούμε, γιατί γυναίκα του ψωνίζει στο Παρίσι. Αλλά τέλος πάντων, ένα χρόνο πριν, τον περασμένο Ιούνιο, α, αν είχαμε πάρει αυτές τις αποφάσεις, νομίζω ότι θα είχαμε αποφύγει το χειρότερο από αυτά που ζούμε σήμερα. Το τραγικό είναι ότι ακόμα και σήμερα δεν είμαστε στο ύψο των περιστάσεων. Δεν θέλουμε να προχωρήσουμε. Γι' αυτό έχω μια ερώτηση προ τον κύριο Μιγκαρέλ. Τι ε, καρότο και μπαστούνι θέλουμε να τραντάξουμε απέναντι στη Ρωσία. Τι μπορούμε να δώσουμε ως κίνητρο. Τι μπορούμε να επιβάλλουμε ως τιμωρία, ως κύρωση. Δεν αρκεί να παραπονιόμαστε για τους Ρώσους. Τι προβλέπουμε να κάνουμε γι' αυτό. Έχω τώρα μια ερώτηση για το πώς θα προχωρήσουμε στα πλαίσια του ΟΗΕ. Η μία εναλλακτική θα ήταν η αναδιατύπωση της εντολής της σημερινής ε, αντιπροσωπείας, της σημερινής αποστολής. Δηλαδή, να γίνει μια πραγματική αποστολή παρατηρητών με βάση το άρθρο 7. Αυτό είναι διαφορετικό από την στρατιωτική παρέμβαση, γιατί ε, ναι, μεν δεν θα ήταν ε, όσοι είναι σήμερα εκατοντάδε, δηλαδή θα ήταν χιλιάδε, αλλά και πάλι δεν είναι στρατιωτική παρέμβαση. Για το θέμα τη ε, ενότητα. Ίσως θα πρέπει να υιοθετήσετε το σύνθημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ενωμένοι μέσα στην διαφωνία μας, μέσα στην πολυφωνία μας. Ίσως σας βολεύει και σας αυτό. Ο κύριος Στάνοκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ με εκείνους που πιστεύουν ότι έχει πεθάνει το, το σχέδιο ε, Ανάν και χρειάζεται να βρούμε κάτι άλλο. Τώρα αυτό το οποίο λέγεται για την ενότητα των αντιπολιτευόμενων και αν θα μπορούσε να εξευρεθεί μια χριστιανική συνιστόσα αλαβητών θα ήταν κάτι ανακουφιστικό. Ακούμε για τον άσταθμο της, ε, στην Ταρτισό και ε, στην και ακούμε και επίσης ε, φήμες ότι παραμένει ο ε, Μπασάρα Λασάντ και ότι ε, ίσως θα έπρεπε να εξεταστεί μια άλλη δυνατότητα ότι κάποιος άλλος θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει στην εξουσία Ποια είναι η δική σας άποψη. Θα ήταν αποδεκτή μια άλλη μορφή συνασπισμού κυβερνητικού με κάποια πλειοψηφία ε, από τον Πάθα και προοπτική δημοκρατικών εκλογών ή όχι. Αληθεύει ότι θα έπρεπε να υπάρξουν δυνάμεις τώρα που όπως ε, καταλαβαίνω είναι ε, συμμορίες ε, αλαβητών και είναι η μόνη αξιόπιστη δύναμη επιβολής της τάξης για τη Δαμασκό μια και οι περισσότεροι στρατιώτες λιποτακτούν και έχουν λιποτακτήσει αληθεύει αυτό η παρουσία της Εσμπολά στην Συρία είναι η επόμενη φάση αυτό θα ζητήσει ο Ασάντ να υπάρξει παρέμβαση, επέμβαση της ε, Χεσμολά για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του. Τι μπορεί να κάνει η Τουρκία. Υπάρχει κάποια ευκαιρία στο Συμβούλιο Συνεργασίας ε, ε, των κρατών του κόλπου, του Περσικού κόλπου να υπάρξει μια προοπτική επέμβαση δράσης της Τουρκίας. Υπήρξε και η δυνατότητα παρέμβασης στο Κόσοβο χωρίς την υποστήριξη του Συμβουλίου ασφαλεία. Και ίσως η άλλη, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση, να υπάρξει μια δυνατότητα να ξεπεράσει ξεπεραστούν ε, τα ε, βέτο της ε, Ρωσίας όσον αφορά την προστασία ειρήνευσης. Είναι μια φαιά ζώνη όσον αφορά τη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει υπό εξέταση μια τέτοια προοπτική και σε σχέση με την ICC που αυτή τη στιγμή υπό τα βέτο της Ρωσίας και της Κίνας έχουν τροχοπεδηθεί. Αν υπήρχε μια στρατιωτική επέμβαση, μια ζώνη ασφάλειας ε, θα ήταν δυνατόν να δημιουργηθεί σε σχέση με εκείνους που θα επέμβαιναν στην ε, Συρία. Ευχαριστώ. Μέιερ. Κύριος Μέιερ. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Μάιερ. Αύριο νομίζω ότι ο στρατηγός ε, κ. Ρόμπερτ που είναι υπεύθυνο ε, για την παρατήρηση, αποστολή παρατήρησης θα εμφανιστεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Οι λόγοι για τους οποίους ζητήθηκε η, ε, η ακύρωση αυτής της αποστολής και οι δύο πλευρές και αναφερόμαστε στην κυβέρνηση του Ασάντ και την αντιπολίτευση κατηγορούνται γιατί δεν έχουν καμία βούληση, είπε, να εξεύρουν μια ειρηνική λύση και κατηγόρησε και τις δύο αυτές πλευρές για δολοφονίες και βιοπραγίες. Θα έπρεπε να υπάρξει κάθε ε, αλληλεγγύη από την ομάδα μας προς, τις, ε, προς τους Σύριους. Δεν αξίζει να έχει τέτοια αντιμετώπιση ο λαός της Συρίας. Ο ίδιος ε, αυτός ο στρατηγός απίθυνε έκκληση προς τα μέρη ώστε να υπάρξει η απομάκρυνση των ηλικιωμένων, των γυναικών, των παιδιών, των τραυματισμένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις εκεί όπου υπάρχουν οι ένοπλες σειράξεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και αντιπολίτευσης. Και πιστεύω ειλικρινά πρέπει να πω τούτων λεχθέντων ότι σε σχέση με αυτούς που λένε ότι πρέπει να υπάρξει μια στρατιωτική επέμβαση όπως στη Λιβύη, εγώ δεν το συμμερίζομαι. Δεν συμμεριζόμουν και του λόγους επέμβαση στη Λιβύη και ούτε συμμερίζομαι να υπάρξει, ούτε μπορώ να συμφωνήσω να υπάρξει μια στρατιωτική επέμβαση επέμβαση στη Συρία. Και γι' αυτό λοιπόν όπως αναφέρθηκε από τον ίδιο του στρατηγό θα πρέπει να ζητηθεί να επιβληθεί και στις δύο πλευρές να εξευρεθεί ειρηνική λύση ώστε να συνέρθουν γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι. Δεν έχει πιστεύω δεν έχει αποβιώσει το σχέδιο Ανάς, Ανάν και χαιρετίζουμε του να, το δημιουργηθεί μια ομάδα επαφής ε, που θα συνέρθει στη Γενέβη όπου θα συμμετάσχει επιπλέον και το ίδιο το Ιράν και αυτό είναι ε, ε, αίτημα του ιδίου του Ανάν όχι της ουσίας για να μπορέσει να ε, αντανακλά τα συμφέροντα όλων που εμπλέκονται σε αυτή την αντιπαράθεση. Να αποφύγουμε τον εμφύλιο πόλεμο και τις σειράξεις. Και σε σχέση με τα όσα είχαν ε, ο Πούτιν και ο Ομπάμα είπαν στη συνάντηση της Λέσχης των 20, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια σημεία συνένεσης μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ για να αναζητηθεί πραγματικά η δυνατότητα μιας προοπτικής πολιτικής επίλυσης του προβλήματος αυτού. Και πιστεύω ότι υπό το δικό μας πρίσμα η λύση πρέπει να είναι πραγματικά πολιτικού χαρακτήρα, πολιτικής φύσης, απευθύνοντας έκκληση στα μέρη και στις δύο πλευρές, όπως και ο ίδιος ο στρατηγός Ρόμπερτ μου το ανέφερε, πρέπει να είναι υπεύθυνοι και οι δύο, και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Και βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη αυτής της βούληψης και γι' αυτό πιστεύω ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να εξετάζουμε μέχρι να εξαντληθεί αυτή η προοπτική, μια τέτοια δυνατότητα. Και από πλευράς λοιπόν του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να πούμε ότι σε σχέση με οποιουσδήποτε εκπροσώπους της κυβέρνησης και του καθεστώτος δεν έχουμε καμία τέτοια συμπάθεια. Αν όμως μπορούμε να συνεισφέρουμε, να συνεχιστεί ο διάλογος και να επιβληθεί ο διάλογος ώστε να εξευρεθεί μια μεταβατική λύση, ειρηνική λύση, αυτό θα μπορούσε να γίνει. Ο κύριος Μπάντα παρακαλώ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι με τον κύριο Μέγερ συμφωνώ απόλυτα. Αν την κλιμάκωση της βίας την δει κανείς, πρέπει να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του κανείς για να εξευρεθεί μια πολιτική λύση σε αυτή τη σύραξη. Θα θέλω όμως να αναφέρω το εξής από άμεσες τηλεφωνικές επαφές και συνδιαλέξεις και ηλεκτρονικά μηνύματα είχα την ευκαιρία με ε, κάποιες τέτοιες επαφές ε, τις τελευταίες εβδομάδες να ακούσω και να μάθω τα εξής. Και θα ήθελα από τους φιλοξενουμένους μας να τοποθετηθούν οι προσκεκλημένοι μας. Άκουσα ότι στο Homs 300 έως 500 περίπου υπερήλικες ηλικιωμένοι και ε, ασθενείς βρίσκονται ως όμοιροι στην ε, εξουσία του καθεστώτος. Είναι τρομακτικό αυτό. Άκουσα επίσης ότι στη Χόμ, στη Χάμα και αλλού υπάρχουν εκατοντάδες χωριά που έχουν ε, με πληθυσμό χριστιανικών μειονοτήτων που από αυτή τη, στιγμή από ε, άτακτες συμμορίες ενόπλων υφίστανται επιθέσεις ε, και πλήττονται, υφίστανται τα πάνδυνα. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας. Αν η ίδια η αντιπολίτευση διαπράττει τέτοια εγκλήματα και φρικαλαιότητες, τότε δεν μπορούμε να επιλέξουμε τον ένα ή τον άλλο, το καθεστώς του Ασάντη ή τους άλλους. Πώς βρίσκεστε εσείς ως αντιπολίτευση, πώς τοποθετήστε έναντι αυτών των ατάκτων συμμοριτών ε, των αντιπολιτευομένων, των ε, αντιφρονούντων που ε, κάνουν τέτοιες επιθέσεις σε αυτά τα χωριά. Είδα πολλές φωτογραφίες τις τελευταίες ημέρες που δείχνουν ότι οι ομάδες ανταρτών επίτηδες έχουν προβεί σε αυτές τις εσκεμμένες βιοπραγίες. Τι γνωρίζετε εσείς θέλω να ρωτήσω για αυτή την κατάσταση της χριστιανικής μειονότητας όπως την περιέγραψα σε αυτά τα χωριά. Και δεύτερη ερώτηση, τι γίνεται με την, Τουρκη... με την κουρδική μειονότητα. Υπάρχουν πολλές μειονότητες μειονότητες και η κουρδική είναι και αυτή μια σημαντική για την αλλαγή στη Σύρια. Θα δώσω το λόγο σε όλους ε, να απαντήσουν και στον ε, κύριο Μιγκαρέλη και στους τρεις εισηγητές μας. Αλλά θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μιγκαρέλη. Ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η θέση της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφάλειας. Και ήθελα να ρωτήσω πόσο σημαντικό ενδιαφέρον ε, πόσο, πόσο, κρίνει, πόσο σημαντικό κρίνει ότι είναι ε, το συμφέρον της Ρωσίας, το πολιτικό και το οικονομικό, κυρίως σαν αφορά το λιμάνι της Τάρτης. Ε, τι θα κάτι είναι πρώτη διατεθειμένη... Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Θα ήθελα να πω τρία πράγματα. Καταρχάς όσον αφορά την ένωση, αν θέλετε, των, των αντιπολιτευομένων. Έχουμε 20 εκατομμύρια που είναι αντίθετα στην, στο καθεστώς και είναι μια αντιπολίτευση η οποία είναι οργανωμένη γεωγραφικά αν θέλετε. Υπάρχει τοπική αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση του εξωτερικού και θα πρέπει να ε, βρούμε στοιχεία κοινά που να ενώνουν την αντιπολίτευση και να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις εξωτερικές παρεμβάσεις. Η Παλαιστινιακή Αρχή έχει, είχε προετοιμάσει μία ε, επίσκεψη στη Ρωσία και πήγα στη Ρωσία και εξήγησα και προσπάθησα να μιλήσω με τους Ρώσους δεν μου είπαν όμως κάτι συγκεκριμένα, απλώς οι Ρώσοι θέλουν να τιμωρήσουν τους Δυτικούς για την παρέμβασή τους στην Λιβύη. Δεν έχουν κάτι συγκεκριμένο με τη Συρία. Ε, θέλουν να αναγκάσουν τους Δυτικούς να βρούνε μια γενικότερη λύση για τα προβλήματα της περιοχής. Δεν έχουν τίποτα για τη Συρία συγκεκριμένο. Και τους ζητήσαμε να μην, ε, να μην χωρίσουν αν θέλετε τη χώρα μας ε, και απλώς θέλουν οι Ρώσοι, επαναλαμβάνω, να πληρώσουν δυτική. Τώρα, για την ε, ειρηνική επίλυση. Εμείς σας είπαμε ότι θέλουμε μια ειρηνική λύση. Ναι, όμως για να βρεθεί η ειρηνική λύση πρέπει να φύγει ο δικτάτορας, πρέπει να φύγει αυτός ο αιμοσταγής ε, ε, δικτάτορας και μετά να εφαρμοστεί το σχέδιο Ανάν μέσω της δημιουργίας μιας, εθνικής, ε, μιας κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας. Και μας είπαν όμως ότι ο Ασάντ δεν φεύγει. Ναι, εμείς λέμε ότι θα πρέπει να ασκηθεί πίεση από τη διεθνή κοινότητα για να φύγει ο Ασάντ και το πιο εύκολο είναι να υποστηριχθεί η εσωτερική αντιπολίτευση έτσι ώστε αυτή η εσωτερική αντιπολίτευση να πιέσει την, για την αποχώρηση του Άσαντ. Διότι για να βρεθεί λύση πρέπει να φύγει η οικογένεια Άσαντ. Πρέπει να γυρίσουμε τη σελίδα. Πρέπει να προετοιμάσουμε την άφηξη ειρηνευτικών δυνάμεων στην περιοχή. Πρέπει να ενισχύσουμε την εσωτερική αντιπολίτευση για να επέλθει μια ισορροπία, διότι το καθεστώς δεν είναι ισχυρό. Πάρα πολλοί στρατιώτες είναι διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν το στρατό. Αρκεί να τους υποσχεθεί κάποιος ότι θα προστατευτεί, θα προστατευτεί η οικογένειά τους. Άρα θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτό το κίνημα, αν θέλετε, να υπάρχουν στρατιώτες οι οποίοι να λιποτακτούν από τον Συριακό στρατό. Και αυτή τη στιγμή προφανώς υπάρχουν και κάποια εγκλήματα, αν θέλετε, τα οποία διαπράττουν και μέλη της ε, ε, αντιπολίτευσης. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το καθεστώς είναι υπεύθυνο για αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, αυτή τη μια κατάσταση παρανομίας εκτός νόμου ε, που έχει δημιουργηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα παρελθόν το οποίο δεν είναι και τόσο μακρινό το περιοδικό Der Spiegel είχε πάρει μια συνέντευξη έναν πρώην Υπουργό Άμυνας και μας είπε ότι καταλάβαμε το καθεστώς με βία, άρα θα το εγκαταλείψουμε πάλι με βία. Αυτή είναι η λογική του καθεστώτος. Οι σφαγές ξεκίνησαν τη δεκαετία του 80. 70.000 οβίδες ε, ε, χτύπησαν τον Συριακό λαό και το καθεστώς παρέμεινε. Σε μια προηγούμενη επίσκεψή μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχα δώσει ένα κατάλογο 200 ατόμων που τους χαρακτήρισα ως δολοφόνους και ζήτησα να τιμωρηθούν. Σήμερα ο κατάλογος Υπάρχει ένας κατάλογος 60 ατόμων ε, που δεν θα πρέπει να τους επιτραπεί να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης συζητήσαμε ε, οι πρέσβεις οι πρέσβεις Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποχωρήσουν από τη Συρία. Η απάντηση ήταν ότι δεν μπορούν οι πρέσβεις να, να, εγκαταλείψουν τη θέση τους. Τελικά το έκαναν, αλλά καθυστερημένα και δεν, ε, δεν είχε κανένα αντίκτυπο η χειρονομία αυτή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα καθεστώς το οποίο είναι σάπιο, είναι σάπιο από τη ρίζα του. Δηλαδή πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα καταρρεύσει όπως η Ρωσία ας πούμε, που ξαφνικά κατέρευσε σαν ένας πύργος από χαρτιά. Ε, κανείς δεν περίμενε να καταρρεύσει η Ένωση και νομίζω ότι το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Το καθεστώς θα καταρρεύσει σαν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα. Ε, το επαναλαμβάνω αυτό. Θα καταρρεύσει αναπάντεχα. Και εάν συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίσετε ένα δίλημα. Πώς θα είναι η, παρέμ... η επέμβαση που θα από την, τον ΟΗΕ, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα, η Ρωσία δεν μπορεί να ασκήσει βέτο και πιστεύουμε ότι θα πρέπει το Διεθνές ε, ε, Ποινικό Δικαστήριο να ασχοληθεί με τα εγκλήματα του καθεστώτος. Κάπου διάβασα ότι το Συριακό καθεστώς νομιμοποίησε τα εγκλήματα και όντως το καθεστώς έχει προσπαθήσει να προστατευθεί από μελλοντικές αποφάσεις του, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Έχω γράψει 8 επιστολές στον Μπασάρα Λάσαντ και έχω στείλει επιστολές σε όλους τους υπουργούς. Τους συνάντησα. Συνάντησα και στρατιωτικούς και κανείς ε, δεν ήθελε να μ' ακούσει. Εδώ και τέσσερα χρόνια λέω στο καθεστώς ότι θα χυθεί αίμα στη Συρία. Πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα στη ρίζα τους. Και όμως τίποτα δεν έγινε. Κανένα πρόβλημα δεν λύθηκε. Επομένως χρειαζόμαστε την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας έτσι ώστε να διώξουμε το καθεστώς αυτό, διότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα διαλόγου ε, με, τον, ε, με το καθεστώς αυτό. Μία είναι η, η προοπτική, η αποπομπή του. Και πραγματικά αισθάνομαι απομονωμένος, διότι τελικά ε, βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί δυτικοί, πολλοί Ευρωπαίοι, οι οποίοι χαιρετίζουν και χαιρετούν τον ε, Λοιπόν, θέλω να μιλήσω για τη θέση της αντιπολίτευσης και τη στρατηγική της για την αλλαγή. Στην αρχή της τρίτης χιλιετίας, όταν πήρε ο Ασάντ Αλασάντ, Μπασάντ Αλασάντ την εξουσία, κληρονομικά από το πατέρα του, ε, στα διάφορα λογοτεχνικά σαλόνια της Δαμασκού μιλούσαμε για τη δικαιοσύνη, για τη μετάβαση, για όλα όσα μπορούσαμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε την κοινωνία μας. Ε, αλλά η απάντηση του καθεστώτος ήταν μαζικές κρατήσεις όλων των ακτιβιστών που υπήρχαν στην ε, κινέζικη σκηνή. Ε, η δημοκρατική αυτή άνοιξη πέθανε πολύ γρήγορα, ήταν θνησιγενής. Και το 2005 είδαμε την άλλη όψη του καθεστώτος Το 2005 έγινε και μια απόπειρα για να προσφύγουμε στο τραπέζι των συζητήσεων για μια δημοκρατική αλλαγή για να αποφύγουμε τον εμφύλιο. Η απάντηση όμως του καθεστώτος ακόμα μια φορά ήταν ξανά μαζικές κρατήσεις του Καμέλα Αλμπουένι του... και άλλων ακτιβιστών που ρίχτηκαν στις φυλακές. Η Συριακή Επανάσταση είδε το φως μόνο όταν η αντιπολίτευσή μας έχασε την ελπίδα ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρξει αλλαγή από το καθεστώς. Στην αρχή της Ιριακής Επανάστασης ήρθε ο Μπασάρα Λασάτ ε, στη συνέλευση για να μιλήσει μίλησε με ύφο πολυμοχαρέ. Αυτό δεν μιλάει στο λαό. Απλώ καταδικάζει τους αντιπάλους του, ε, τους δολοφονεί, τους ρίχνει στι φυλακέ. Τι διάλογο μπορούμε να έχουμε αυτόν τον άνθρωπο. Οι Αλαουίτες επίσης δεν είναι στην εξουσία ε, στη Συρία. Το Μπαθ δεν είναι στην εξουσία. Ο Μπασάρ είναι στην εξουσία. Η οικογένεια του Ασάντ είναι στην εξουσία. Ε, ο πατέρας του Μπασάρ δεν έδωσε την εξουσία σε κανένα παρά μόνο στο γιο του. Το πρόβλημα δεν το έχουμε με τους Αλεουίτες, με τους, χριστιανές, με τους χριστιανούς, με, τους, με τον Μπαθ, το κόμμα του Μπαθ, με άλλες μειονότητες θρησκευτικέ. Δεν πρόκειται για πολιτικές ε, συγκρούσεις, ιδεολογικές συγκρούσεις, ανθρωπιστικές συγκρούσεις ή οτιδήποτε άλλο. Κάνουμε μια επανάσταση για να επιβιώσουμε έχουμε μια απόλυτη αντίθεση με το καθεστώς τη της Συρίας. Το θέμα δεν είναι ποιε μειονότητε έχουμε, δεν είναι τι σκεφτικές πεπιθήσει έχουμε. πολεμάμε για να επιβιώσουμε στη Συρία. Αυτό είναι όλο. Το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η Συρία σήμερα οφείλεται σε παραβιάσεις σοβαρότατες που κάνει το καθεστώς καθημερινά. Μιλάμε για ένα καθεστώς εγκληματιών που ρίχνουν στις φυλακές ε, οποιονδήποτε αντιφρονούντα. Ο κύριος Μιγκαρέλη για να απαντήσει στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Δύο ερωτήσεις κυρίας Μπραντνερ. Αν είναι σόφρον να επιβάλλουμε βαθμιές ε, κυρώσεις. και να γλιτώσει ο Ασάντ καταρχήν και κάποια μέλη της οικογένειάς του. Ε, νομίζω ότι μετά από όσα έγιναν ε, και εκ των υστέρων, κάναμε λάθος, μπορούμε να το πούμε αυτό. Γενικά τα κράτη-μέλη τα οποία μας δίνουν τον κατάλογο των ατόμων και των επιχειρήσεων που θα είναι θύματα των κυρώσεων θεωρούν ότι είναι προτιμότερο να δράσουμε βαθμία, να αυξάνουμε την πίεση λίγο-λίγο, ούτω ώστε να αλλάξει το καθεστώ τη θέση του, παρά να πάμε, ας πούμε, με τοπικά και να επιβάλλουμε τι κυρώσει. Ε, αλλά η εμπειρία έδειξε ότι εμεί είχαμε λάθο και εσεί είχατε δίκιο. Τώρα, πώ να αντιμετωπίσουμε τη Ρωσία. Είναι και το ερώτημα του κυρίου Προβέρα. Νομίζω ότι πρέπει καταρχάς να πείσουμε τη Ρωσία ότι θα έχει ρόλο ε, σε όλη αυτή τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης. Πρέπει να τους καθησυχάσουμε τους ρόλους, ότι σε αυτή την πολιτική μετάβαση από την οποία θα περάσει η Συρία, αυτοί θα έχουν κάποιο ρόλο. Δεύτερον, θα πρέπει να τους πείσουμε ότι τα συμφέροντά τους πολιτικά και οικονομικά στην περιοχή θα λαμβάνονται υπόψη και στο μέλλον και κατά τη διάρκεια της μετάβασης. Τρίτον, θα πρέπει να τους εξηγήσουμε ότι αν συνεχίσουν να υποστρίζουν ένα αναξιόπιστο και καταδικασμένο πια καθεστώς, γιατί πια το καθεστώς Ασάντ είναι καταδικασμένο, νομίζω ότι θα χάσουν οποιαδήποτε αξιοπιστία απέναντι στον αραβικό κόσμο. Το λιμάνι της ε, Τασό, ε, εκεί βρίσκονται τα συμφέροντά τους. Εγώ δεν είμαι στρατιωτικός επαΐων. Εγώ από τη διάβασα όμως δεν έχει τεράστιο, δεν έχουν δεν εστιάζουν εκεί τεράστια στρατιωτικά συμφέροντα. Αυτά μας λέει στρατιωτική πάντως, δεν είμαι εγώ εμπειρογνώμονας. Το, το ενδιαφέρον για αυτό το λιμάνι από πλευράς Ρωσίας είναι περιορισμένο. Μπέλντερ. Διώκονται οι Κούρδοι και οι Χριστιανοί. Σας λέω με βεβαιότητα ότι είναι πολύ ανήσυχοι και οι ΜΕΝ και οι ΔΕ για την περίοδο μετά του Ασάντ. Αλλά σήμερα δεν μπορώ να σας πω ότι σήμερα διώκονται είτε Χριστιανοί είτε Κούρδοι. Δεν λέω ότι δεν συμβαίνει, λέω ότι δεν έχουμε αποδείξεις ότι οι χριστιανοί και οι Κούρδοι στη Συρία σήμερα είναι αντικείμενο διώξεων. Δεύτερος όμιλος. Ρομέρο Λόπες. Για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ερώτησή μου είναι επιμένοντας και εμένοντας σε αυτή την προοπτική για τους παρόντες εδώ από την αντιπολίτευση που τους χαιρετίζω εδώ και θέλω να επιμείνω. Πραγματικά υπάρχει μια στρατηγική της αντιπολίτευσης ως στρατηγική, αυθεντική στρατηγική που θα είναι ικανή να οδηγήσει στο να αποφευθεί ο πόλεμος Κάποιος από εσάς είπε ότι στην κοινή πλατφόρμα συμφωνείτε, ότι στις βασικές θεμελιώδεις αρχές συμφωνείτε για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Συρία. Όμως, ποια είναι η δύναμη εκείνη που είναι πιο σημαντική στην αντιπολίτευση, η πιο σημαντική δύναμη της αντιπολίτευσης που τώρα μπορεί να επιβάλλει μια κοινή στρατηγική αυτό θέλουμε να δούμε. Να υπάρχει μια στρατηγική για να μπορούμε εμεί να συνοδέψουμε αυτή τη στρατηγική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη. Να ξέρουμε αυτή τη στρατηγική για να μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Σε ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο πρώτος γύρος για τις απαντήσεις ε, φώτισε κάποια πράγματα θα πρέπει, και αυτό το είπε ο κύριος Λαβάνη, 20.000 άνθρωποι δολοφονήθηκαν. Άλλοι άπειροι ε, έχουν, διαμελιστεί, έχουν ακροτηριαστεί, έχουν τραυματιστεί, άλλοι βρίσκονται στις φυλακές και όταν λέγεται ότι θέλουμε να έχουμε διαπραγματεύσεις μπορεί να είναι γενναίο αλλά δεν πιστεύω ότι θα δώσει, δώσει κάποιο αποτέλεσμα αυτή η διαπραγμάτευση. Δεν θα δώσει κανένα αποτέλεσμα. Μόνο νεκρός μπορεί να αποτελέσει να, απο, να φύγει από αυτή τη χώρα ο Ασάντ ή ως νικητής να επιβάλλει την εξουσία του. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη λύση. Δεν επέζησε ο Τσαουσέσκου. Να δείτε τι έγινε στη Λιβύη για να δείτε τι μπορεί να γίνει με τον Ασάντ. Για το, στο ποινικό δικαστήριο αν θα πήγαινε θα τον φυλάκιζαν η ισόβια. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια άλλη πρόπτικη και για το σύνολο της οικογένειάς του και της κλίκας του. Λοιπόν, πόλεμος ε, με δυνάμεις εξωτερικού δεν θα μπορέσει να κερδιθεί. Έχουμε σήμερα ήδη εμφύλιο πόλεμο και πόλεμο σπίτι με σπίτι στις σειράξεις ε, στα, στις πόλεις. Ε. Μια συγκεκριμένη ερώτηση έχω. Αν πιστέψει κανείς τις φήμες και τις, ε, τις διάφορες πληροφορίες και σύμφωνα με το CIA έχει τεράστιες αποθήκες και μάλιστα ε, διάσπαρτες σε όλη την επικράτεια της ε, Συρίας με χημικά όπλα. Και τι θα γίνει αν τώρα ανατραπεί ο Ασάντ. Είναι θέμα χρόνου για να ανατραπεί. Ας ρίξουμε μια ματιά στην ιστορία για να καταλάβουμε. Μπορείτε να έχετε τον έλεγχο λοιπόν αυτών των χημικών όπλων ώστε να μην περάσουν στα χέρια άλλων τρομοκρατών όπως της Αλκάιντα ή άλλων τρομοκρατών παραπέρα πέρα από την Αλκάιντα και να, τα, να μην τα χρησιμοποιήσουν αυτοί ε, τήρησα το χρόνο που είχα ως αγορητής, πράγμα που δεν το κάνουν όλοι δυστυχώς εδώ. Ευχαριστώ. Έλαν παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου και την βαθιά ανησυχία μου για τις εξελίξεις στη Συρία. Αναφέρθηκε ότι η ελευθερία δεν μπορεί να επιτευχθεί με μιας. Αναφέρατε το παράδειγμα της Σοβιετικής Ένωσης. Εγώ από εκεί προερχόμαι και σας βεβαιώνω ότι οποιαδήποτε δικτατορία τελικά θα καταρρεύσει. Στο μεταξύ όμως και η αντιπολίτευση είναι καταδικασμένη να συνεργαστεί. Μας ε, καλείται να υποστηρίξουμε την εσωτερική αντιπολίτευση. Το ερώτημα είναι ποιο να υποστηρίξουμε. Πώς να σας υποστηρίξουμε. Με ποια μέσα. Συμφωνώ λοιπόν με τον, με τον κύριο Μιγκαρέλη που σας ζητάει να δημιουργήσετε μια κοινή πολιτική πλατφόρμα που να μιλάει για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Αυτή η πλατφόρμα θα μπορούσε να είναι η βάση αυτής. Το ερώτημα είναι το σημερινό σύνταγμα μπορεί να είναι η βάση για την μελλοντική Συρία. Πρέπει να αλλάξει, πρέπει να τροποποιηθεί. Και μπορεί να υπάρξει μια μη θεοκρατική δημοκρατία στη Συρία μια κοσμική δημοκρατία. Για τη Ρωσία τώρα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ρωσία συνεχίζει να πουλάει υψηλή α, στρατιωτική τεχνολογία, πολεμικά αεροπλάνα στη Συρία. Ξέρουμε επίσης ότι διαβεβαιώνουν τους πολιτικούς παρατηρητές ότι αυτά τα όπλα δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά της αντιπολίτευσης. Εσείς τι γνώμη έχετε χρησιμοποιούνται αυτά τα όπλα κατά της αντιπολίτευσης. Η κυρία Κοπά. Μετά από αυτά που είπε ο κύριος Κέλλον, θα να κάνω εγώ ένα σχόλιο για τη Ρωσία. Σήμερα ε, το ε, Foreign Office της Βρετανίας εξέδωσε ένα ανακοινοθέν για ε, ρωσικά αεροπλάνα που κατευθύνονται προς τη Συρία και αεροπλανοφόρα θα, υπάρξει αντίδραση αν, γίνει αυτή, αν συμβεί κάτι τέτοιο. Επίσης, θέλω και εγώ να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς τη Συριακή Αντιπολίτευση. Η διεθνής κοινότητα βρίσκεται σε αδιέξοδο. Από τη μία πρέπει να παραδεχτούμε ότι το σχέδιο είναι νεκρό και δεν μπορεί να αναστηθεί. Και από την άλλη και αυτό είναι η θέση την, της πολιτικής μου ομάδας των σοσιαλιστών, η πολιτική παρέμβαση στην ε, περιοχή δεν είναι επιθεμητή. Είναι μεγάλος ο κίνδυνος για την περιοχή, για τη χώρα, για τον πληθυσμό, αλλά και την ε, διεθνή ειρήνη στην περιοχή. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τη Λιβύη την κατάσταση. Ε, παρότι ήταν πιο εύκολη υπόθεση η Συρία, παρόλα αυτά έχουμε αντιμετωπίσει με σήμα τις ε, επιπτώσεις ε, επίσης υπάρχει μια ψυχολογική πίεση από τους Ευρωπαίους, γιατί όταν κάθε βράδυ βλέπεις ε, νεκρά παιδιά στην ε, τηλεόραση, αυτό είναι πίεση της κοινή γνώμη για παρέμβαση. Αλλά πιστεύουμε ότι η στρατιωτική λύση δεν είναι σωστή. Θα ήθελα να μου πείτε τι άποψη έχετε για όλα αυτά τα θέματα. Για αυτό το θέμα το συγκεκριμένο δηλαδή. Η κυρία Ντεκέιζερ, τελευταία ομιλητρία και τελευταία ερώτηση που θα ακούσουμε από αυτήν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι σε, την, σε αυτό το σώμα όλοι έχουμε τα ίδια συναισθήματα απέναντι στον Μπασάλα Σαντ. Το θέμα είναι πώς θα τον διώξουμε. Είτε θα συνεχίσει και θα γίνει ένας φρικόδης ε, φίλιος ή θα σκοτωθεί κάπου ή θα καταφέρουμε να διαπραγματευτούμε την αποχώρησή του. Δεν βλέπω άλλη λύση. Εσείς είσαστε γνωστοί αντιφρονούντες, σας γνωρίζω, σας χαιρετίζω και τους τρεις. Ειδικά τους δύο που δεν βλέπω εδώ στο Κοινοβούλιο για πρώτη φορά. Και έχετε δείξει εδώ και πολύ καιρό την αποφασιστικότητά σας. Όταν σας ακούμε, θέλουμε πραγματικά να σας βοηθήσουμε. Αλλά όπως είπαν και οι συνάδελφοί μου, δεν ξέρω πώς να το κάνουμε. Λέτε, υποστηρίξτε την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση, εντάξει, την ακούμε, βλέπουμε. Βλέπουμε όμως και όλους αυτούς τους νέους στη χώρα που εξεγείρονται και που είναι διάδοχοί σας. δεν ξέρω όμως πώς να τους βοηθήσουμε. Ξέρετε πολύ καλά τι άποψη έχει το Κατάρι, η Σαουδική Αραβία ε, και τα όπλα που στέλνουν. Ε, κυκλοφορούν πολλά όπλα. Δεν είναι όπλα αυτό που θέλουμε να τους δώσουμε. Ε, τώρα, νομίζω αν κάνουμε στρατιωτική παρέμβαση θα, πως αποσταθεροποιούσαμε την ε, περιοχή. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν εμείς. Πέρα από την άσκηση πολιτικών πιέσεων και διαπραγματεύσαμε τη Ρωσία, ούτω ώστε η υποστήριξη της Ρωσίας απέναντι στον Μπασάρα Λασάρ να σταματήσει και να δικαστεί και να διωχθεί με κάποιο τρόπο. Πέρα από αυτό που σας λέω, δεν μπορώ. Τι, μπορώ να σας, πω, τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να σας βοηθήσω με τρόπο που να μην είναι καταστροφικό για εσάς και τη χώρα σας. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο για τις απαντήσεις βέβαια, δυστυχώς. Σύντομες απαντήσεις σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Το μεταβατικό σχέδιο θα ξεκινήσει με την αναχώρηση του Άσαντ και η εφαρμογή του σχεδίου Ανάν στο σύνολό του και η δημιουργία ενός νέου συντάγματος μπορούν μόνο να ξεκινήσουν μόνο εάν φύγει ο Αλ Άσαντ. Πρέπει να υποστηρίξουμε τον λαό της Συρίας. Έχουμε και άλλους φίλους που μας υποστηρίζουν. Εμείς, από Σάσα χρειαζόμαστε διπλωματική βοήθεια. Και εσείς πρέπει αυτό το να ε, συνεχίσετε να κάνετε διπλωματική υποστήριξη. Ο Ελάσαντα πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στην αποχώρηση στο θάνατο. Φαντάζομαι ότι θα διαλέξει την αποχώρηση. Επίσης υπάρχουν πολλές ομάδες, πολλές συμμορίες που έχει οργανώσει το ίδιο το καθεστώς που, ε, που τους έχει δώσει όπλα και που διαπράττουν διάφορα εγκλήματα. Αυτό το οποίο θέλουμε εμείς είναι να βρεθεί μία ειρηνική λύση, έτσι ώστε και οι προσπάθειές μας να στεφθούν με επιτυχία. Κοιτάξτε, από την πλευρά μου πιστεύω ότι η έκθεση του ΟΗΕ, η έκθεση που λέει ότι 3 εκατομμύρια Σύριοι χρειάζονται βοήθεια, πιστεύω ότι μιλάμε για πολύ μικρό αριθμό ατόμων. Όσα, τα χρήματα, όσα χρήματα έχουν δοθεί μέχρι τώρα δεν αρκούν η Τουρκία είχε, είχε δηλώσει την θέλησή της να οργανώσει ένα διεθνές συνέδριο για να ε, βοηθήσουν τον λαό της Συρίας. Αυτό το οποίο λέω εγώ είναι ότι θα πρέπει καταρχάς να υπάρχει και να συνεχίσει να υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια και κατά δεύτερον να πιστεί το καθεστώς να αφήσει ελεύθερη την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας γιατί αυτή τη στιγμή σταγόνα σταγόνα μπαίνει η ανθρωπιστική βοήθεια. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει με το στρατό διότι 3.000 άρματα έχουν κυκλοφορούν ε, από πλευρά τη κυβέρνηση Για να μην μιλήσω για τους βόμβε, για τι οβίδε, για τι χειροβομβίδε, για τα... δεν ξέρω κι εγώ και τι άλλο. Δεν, μπορεί, να, μπορεί να πει κανείς ε, ότι υπάρχει ε, ισορροπία δυνάμεων και όταν ζητάμε κατάπαυση πυρός τι σημαίνει Πώς μπορεί να υπάρξει κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε έναν στρατό ο οποίος είναι οπλισμένος και στον λαό που δεν είναι οπλισμένος, που είναι άοπλος. Είναι ένα ψέμα επομένως όταν μιλάμε για κατάπαυση πυρός. Παρά τις διαφορές μας υπάρχει μια μακραίωνη αν θέλετε ιστορία φιλίας ε, και πρέπει στην περιοχή να υπάρξουν καθεστώτα τα οποία να είναι δημοκρατικά, να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελπίζω και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι αρρωγός στις προσπάθειές μας. Επίσης ε, για το μποϊκοτάρισμα και την απομόνωση του καθεστώτος πιστεύω ότι είναι καλά μέτρα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν δύο πρακτικές λύσεις. Αυξημένη πίεση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη, Ρωσία στα πλαίσια του Συμβουλίου Ασφαλείας, ούτως ώστε να περάσει ένα ψήφισμα που στο πρώτο σημείο θα απαιτεί την αποχώρηση του Μπασάρ Λασάντ και την προσαγωγή του στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε επίσης, να βοηθήσετε τους ακτιβιστές, να εξασφαλίσετε την ασφάλειά τους, ειδικά όταν κάνουν διαδηλώσεις και πορείες. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης και κάλυψη από τα ΜΜΕ που απαγορευόταν μέχρι μέχρι τώρα. Ε, υπάρχουν ε, ακτιβιστές που έχουν πάει στην Ιορδανία, στην Τουρκία, ε, γιατί απειλείται η ζωή τους, θα πρέπει να βοηθηθούν και ζητάμε περισσότερη βοήθεια από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε αυτούς τους ακτιβιστές που έχουν καταφύγει σε διάφορες χώρες, γιατί κινδυνεύει η ζωή τους. Να κάποιες πρακτικές λύσεις που μπορείτε να βοηθήσετε και να περάσατε. Ευχαριστούμε πάντως ειλικρινά την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλη τη βοήθεια που έχει δώσει σε αυτόν τον τομέα. Θα πρέπει να φτάσουμε σε μια γρήγορη λύση και να απειλήσουμε απερίφραστα τον Μπασάρ Λασάντ. Πρέπει να τον εξαναγκάσουμε να παραιτηθεί. Ακόμα και αν δεν υπάρχει ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, Ακόμα και αν δεν βομβαρδίσουμε, <laughs> ε, θα πρέπει τουλάχιστον να τον αναγκάσει να φύγει. Κύριος Μιγκαρέλη, ε, εμείς δεν θέλουμε να υπάρξει στατικοποίηση της σύγκρουσης ε, και δεν συμφωνούμε με άλλους. Υπάρχουν άλλοι που συμφωνούν, που τη θέλουν. Ε, πάντως αυτή είναι μία θέση, καταρχάς, έτσι που παίρνουμε. Δεύτερον, η έχουμε θετήσει ένα εμπάρκο όπλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητήσαμε από όλου του ενδιαφερόμενου, του εμπλεκόμενου και κυρίω τη Ρωσία να σταματήσει να χορηγεί όπλα στο καθεστώ Ασάντ. Τρίτον, δουλεύουμε αυτή τη στιγμή ούτω ώστε οι κυρώσει μα να μπορέσουν να εμποδίσουν ε, την παράδοση των όπλων. Ζητάμε, ας πούμε, στις ευρωπαϊκές εταιρείες να μην εξασφαλίσουν ε, βρίσκουν τα όπλα τα οποία μεταφέρουν τα, συγγνώμη, τα σκάφη που μεταφέρουν τα όπλα προς τη Συρία. Ε, δουλεύουμε με τα κράτη-μέλη για αυτό το θέμα ήδη αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία, μακρά η συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ τους εισηγητές και τους ομιλητές. Καλή τύχη για σας προσωπικά και για τη χώρα σας. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστώ τον κύριο Μιγκαρέλ που ήταν πάντα ε, πολύ συγκεκριμένος. Σας ευχαριστώ όλους.